Dear colleagues, it is time to start to vote. Now we can go to the item 9 in our agenda. Περνάμε στο σημείο 9 της ημέρης της διάταξης, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά την, για την προφορική ερώτηση που αφορά την απόφαση της Ιαπωνίας να συνεχίσει τη φαραναθυρία κατά την περίοδο 2015-2016, την ελληνική περίοδο. Αν έχετε φέρει τις κάρτες, τις ηλεκτρονικές κάρτες ψηφοφορίας, μπορείτε να ψηφίσετε. Άχρη ψηφοφορία. Okay.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 να κλείσουμε την ψηφοφορία. Εντάξει, εντάξει. Εγκρίνεται. Πανψηφί. Περνάμε στο δεύτερο. Στο δεύτερο θέμα για ψηφοφορία. Question to the Council. Ερώτηση προς το Συμβούλιο. Everybody have voted. Ψηφίσατε όλοι. Εγκρίνεται. Επόμενο σημείο της σημερινής διάταξης μετά τις ψηφοφορίες είναι το σημείο 10 έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την εφαρμογή της απόφασης για τις σοβαρές διασυνοριακές απειλές ε, κατά της υγείας και την κατάργηση της απόφασης 2119. Θα ακούσουμε πρώτα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον κύριο Τζον Ράιον, ε, που ασχολείται με τα θέματα της ε, διαχείρισης κρίσεων στην Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΤΕ. Παρακαλώ όσοι θα φύγουν από την αίθουσα να το κάνουν γρήγορα και αθόρυβα για να δώσουμε την ευκαιρία στον κύριο Ράιαν για να μας εξηγήσει τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 19 της απόφασης και που προβλέπει υποβολή της έκθεσης ήδη από πέρυσι τον Νοέμβριο. Διακόπτει ο πρόεδρος. Συνεχίστε. Και κάθε τριετία. Αυτή είναι η πρώτη λοιπόν έκθεση από μια σειρά εξέσεων που σκοπό έχουν την αναθεώρηση της απόφασης. Σε ό,τι αφορά το ιστορικό υπόβαθρο, η απόφαση αυτή 1082 του 2013 αντικαθιστά προηγούμενη απόφαση νομοθετική πρόταση που ίσχυε για πολλά χρόνια και που αφορούσε μόνο τις μεταδοτικές ασθένειες μετά το ξέσπασμα του SARS. Οπότε η αλλαγή του νέου κειμένου σχέση με το παλιό είναι ότι διευρύνει την κάλυψη ε, του συστήματος από τις μεταδοτικές μονονόσους προς όλες τις απειλές. Καλύπτει και τις περιβαλλοντικές απειλές και τις απειλές βιοτρομοκρατίας. Οπότε διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής της απόφασης αυτή τη φορά. Το πρώτο βασικό επίτευγμα της νέας νομοθεσίας είναι η ε, επισημοποίηση της Επιτροπής ε, Υγείας και Ασφάλειας που συστήθηκε από το Συμβούλιο του 2001 σε άτυπο επίπεδο, σαν επίσημο και το, ε, η απόφαση 1082 του 2013 επισημοποιεί την Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας που επιτρέπει στα κράτη-μέλη να συντονίζονται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον τρόπο που θα ανταποκριθούν στις διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας. Άλλο ενδιαφέρον στοιχείο της νέας νομοθεσίας που περιλαμβάνεται στο σημείο στη σελίδα 4 της έκθεσης αφορά την ετοιμότητα για την αντιμετώπιση σοβαρών διασυνοριακών απειλών. Εδώ έχουμε και πάλι ε, επέκταση του πεδίου εφαρμογής καλύπτει και η ετοιμότητα. Τα κράτη-μέλη δηλαδή είναι ε, υποχρεωμένα να είναι σε ετοιμότητα για να αντιμετωπίσουν τέτοιες σοβαρές διασυνοριακές ε, απειλές και να ενημερώνουν τακτικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πώς έχουν εφαρμόσει τις συστάσεις των διεθνών δεταξιών και συντονισμού του τομέα της υγείας με άλλους τομείς και εξασφάλιση μια συνέχεια. Αυτό είναι το δεύτερο λοιπόν στοιχείο της νέας απόφασης. Έχουμε μια νέα Επιτροπή ασφάλεια και προστασία και ενισχύεται η έκθεση ώστε να περιλαμβάνει και την ετοιμότητα. Κάνουμε και την πρώτη επισκόπηση, την πρώτη έρευνα στα κράτη-μέλη για να δούμε πόσο έχουν αυξήσει την ετοιμότητά του να αντιμετωπίσουν τέτοιε σοβαρέ διασυνοριακέ απειλέ. Αυτό είναι το αντικείμενο τη έκθεση που εξετάζουμε τώρα στην Επιτροπή Ασφάλεια και Υγεία εντοπίστηκαν κάποια προβλήματα, κάποιες αδυναμίες στην έκθεση και προσπαθούμε με τα κράτη-μέλη να τα διορθώσουμε. Για παράδειγμα, ανάπτυξη ασκήσεων με τις επενδύσεις από το πρόγραμμα υγείας στις αξιολογήσεις αναχώρα. Έχουμε διάφορες πρωτοβουλίες κατά νου, ανάλογα με την αξιολόγηση που θα γίνει ε, των διαφόρων ε, ασθενειών και το ξεσπάσματος για να ενισχύσουν την ετοιμότητα στα κράτη-μέλη. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα μέτρα αντιμετώπιση. Αυτό είναι ένα νέο στοιχείο της ε, νέας νομοθεσίας. Τα κράτη-μέλη μπορούν να θεσπίσουν από κοινού κάποια μέτρα για να αντιμετωπίσουν μεταδοτικές νόσους και ευτυχώς έχουμε ήδη την υπογραφή από 14 κράτη-μέλη που ήδη στις 20 Ιουνίου του 2014 είχαν υπογράψει και πλέον νέα, ε, νέα, νέα κράτη ε, συνυπέγραψαν. Και η, η συμφωνία για τις κοινέ ε, συμβάσεις έχει προχωρήσει και τον Απρίλιο Ελπίζουμε και η Γερμανία να προσυπογράψει τη συμφωνία. Κάτι που σημαίνει ότι έχουμε συγκεντρώσει μεγάλο αριθμό κρατών μελών που έχουν ήδη υπογράψει αυτή τη δυνατότητα να αγοράσουν από κοινού, να ε, υιοθετήσουν από κοινού τέτοια μέτρα. Αρνητική μέχρι στιγμή ήταν η απάντηση μόνο από τη Βουλγαρία και την Πολωνία. Μόνο αυτές ε, οι χώρες δεν έχουν συμμετέχει μέχρι στιγμή σε αυτές τις κοινέ ε, προσπάθειες σε ό,τι αφορά την επιδημιολογική επαγρύπνιση και παρακολούθηση, η συγκέντρωση στοιχείων για ε, ασθένειες, ε, για ξέσπασμα ασθενειών και ε, επαγρύπνηση. Για να σας δώσω μία ιδέα, έχουμε 47 νόσους που καλύπτονται από το σύστημα. Και όταν ε, έχουμε εμφανίσει τέτοιων κρούσματα τέτοιων ασθενειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη-μέλη υποχρεούνται να κοινοποιήσουν στο κοινοτικό σύστημα και συναγερμού για τα κρούσματα, αλλά και ε, στατιστικά στοιχεία για αυτές τις 47 νόσους. Επιπλέον, από την επίσημη αυτή απόφαση, έχουμε και ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης. Ένα πιστευτικό ηλεκτρονικό σύστημα που επιτρέπει στα κράτη-μέλη να ανταλλάξουν πληροφορίες για κρούσματα νόσων. Και αυτό χρησιμοποιείται καθημερινά. Και μάλιστα στη σελίδα 8 της έκθεσης βλέπετε είχαμε 168 μηνύματα. Και 354 σχόλια. Βλέπετε είναι ένα πολύ ε, ζωντανό σύστημα που επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών για κρούσματα. Και μάλιστα σήμερα είχαμε την ειδοποίηση για ένα κρούσμα ε, ψηλού πυρετού και μάλιστα με τον ιό Ζήκα πολλά ε, μηνύματα κυκλοφόρησαν μέσω του συστήματος και στο, στην 8, στη σελίδα 8 βλέπετε ε, ποια είναι τα μηνύματα και για ποιες ασθένειες, από ποιες χώρες και για ποιες, σε ποιες ασθένειες αναφέρονται. Επίσης, έχουμε και εκθέσεις αξιολόγηση κινδύνου που αποτελούν τη βάση για τα μέτρα συντονισμού που λαμβάνουν τα κράτη-μέλη και βλέπετε στην έκθεση ότι είχαμε 28 αξιολογήσεις κινδύνου την περίοδο από το κέντρο ε, της πρόληψης ε, νόσων και συναντήσεις για να εξετάσουμε αυτές τις αξιολογήσεις κινδύνου. Επίσης, ε, με βάση την νομοθεσία αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να κηρύξει έκτακτη ε, υγειονομική ανάγκη. Κάτι που δεν έχει χρησιμοποιηθεί ακόμη γιατί το έχει κάνει στη θέση μας η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Για την πολιομελίτιδα, για το έμπολα και τώρα για τον ιό Ζήκα. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας ήταν αυτή που κήρυξε έκτακτη υγειονομική ε, κατάσταση. Οπότε δεν χρειάστηκε να ασκήσουμε εμεί αυτή τη δυνατότητα ω Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πάντω η έκθεση κάνει γενικώ μια καλή επισκόπηση για τον τρόπο εφαρμογή απόφαση από την έγκρισή τη. και πρόκειται για ένα κινούμενο στόχο, γιατί κάθε μέρα ουσιαστικά έχουμε ένα νέο κρούσμα, μια νέα αρρώστια, νέα αξιολόγηση κινδύνου, νέα μέτρα που χρειάζεται να ληφθούν. Οπότε πολλέ από τι πληροφορίε αυτέ δείχνουν απλώ ένα στιγμιότυπο μια δεδομένη στιγμή, γιατί από την δημοσίευση της έκθεσης και μετά πολλές εξελίξεις είχαμε. Αυτά, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και να δώσουμε το λόγο παρά αυτά. Στον ε, πρώην εισηγητή για τέτοια θέματα, ο κ. Παρνιό ήταν ο προηγούμενος εισηγητής. D'abord, euh, comme vous venez de le rappeler euh, j'ai été σας ευχαριστώ να σας πω ότι όντως ήμουν εισηγητής για την ε, αποφάσεις για τις διασυνοριακές απειλές προς την υγεία στην προηγούμενη θητεία. Και θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω το Γενικό Γραμματέα της ε, Γενικής Διεύθυνσης ε, Υγείας που μας έκανε την παρουσίαση του αυτή πολύ ωφέλιμη για το κείμενο αυτό. Να σας πω ότι όχι μόνο συνεργαστήκαμε καλά για την προετοιμασία του κειμένου και να ευχαριστήσω τον Τζον Ράιεν, ο οποίος ε, συνέχισε να με ενημερώνει και μετά τον ε, πρώτο απολογισμό και έτσι μου επέτρεψε ως Ευρωβουλευτή να δω ότι πραγματικά υπήρξε συγκεκριμένη εφαρμογή των όσων αποφασίσαμε εδώ. 6 Νοεμβρίου του 2013 λοιπόν ε, τέθηκε σε εφαρμογή η απόφαση αυτή για την προστασία της υγείας των Ευρωπαίων από μεταδιδόμενες νόσους και από τις διασυνοριακές αυτές απειλές, όπως είπατε, ο μηχανισμός ε, αυτός δοκιμάστηκε άμεσα από την επιδημία του εμπόλα που άγγιξε την Δυτική Αφρική το Μάρτιο του 2014 μέχρι τον ε, Ιανουαρίο του 2016 28.600 άτομα ε, νόσησαν στην Αφρική και 11.311 έχασαν τη ζωή του. Τότε η διεθνή κοινότητα ε, αντέδρασε με μεγάλη καθυστέρηση και νομίζω, ε, μάλλον μιλάω για την Διεθνή Επιτροπή Υγείας και όχι για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ λοιπόν στην Επιτροπή μας ε, σε ό,τι αφορά τον εμπόλα διαπιστώσαμε ότι η τα ευρωπαϊκά μέτρα τα οποία εφαρμόστηκαν μας επέτρεψαν πραγματικά να υπάρξει προστασία στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Και θα πρέπει να εξαγάγουμε λοιπόν τα διδάγματα από τις κρίσεις αυτές της ε, κρίσεις της υγείας και σε ό,τι αφορά τον ε, Δεν θα πρέπει να περιοριστούμε λοιπόν σε μια ανταλλαγή πληροφοριών απλά, όπως έγινε με την περίπτωση του έμπολα, αλλά θα πρέπει πραγματικά να συντονίσουμε την αντιδρασή μας και στο σημείο λοιπόν αυτή, η απόφαση μας, η απόφαση αυτή έχει μια προσθέμενη αξία. Για να ολοκληρώσω αυτή την παρέμβαση, θα ήθελα να απευθύνω μια ερώτηση προς εσάς. Μας είπατε ότι οι πληροφορίες που σας χορηγούν τα κράτη-μέλη στο website EU Survey δείχνουν ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές σε ό,τι αφορά και το σχεδιασμό αλλά και τη συνεργασία μεταξύ των διάφορων τομέων της υγείας. Πείτε μας λοιπόν τι μέτρα ελήφθησαν για να γεφυρώσουν τα χάσματα που εντοπίστηκαν μεταξύ των κρατών μελών. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν και να σας ευχαρώ για την ε, ενεργή δουλειά που κάνατε από το 2013 σε ό,τι αφορά και τα φάρμακα, τα εμβόλια, την αγορά ε, των στοιχείων προστασίας του εξοπλισμού προστασία και στην περίπτωση τη γρήπη. Είδαμε τα κράτη-μέλη, τα οποία δεν είχαν συντονίσει τι δράσει τους, δεν είχαν αγοράσει ενδεχομένω ε, ε, εμβόλια και τελικά τα αποτελέσματα. Βλέπουμε λοιπόν ότι πλέον υπάρχουν κοινά μέτρα, κοινό συντονισμό και αυτό να επενθυμίσουμε ότι οφείλεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, η κυρία Γκροστέκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ για τις πληροφορίες που μας δώσατε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλαδή. Είναι πολύ σημαντικά αυτά με την ε, εξάπλωση ασθενειών όπως τον Ιωέμπολα, τον Ιωζίκα, αυτή τη στιγμή μπορεί να προκύψει και μια οποιαδήποτε άλλη επιδημία ανά πάσα στιγμή. Είναι σημαντικό λοιπόν να μπορούμε να εντοπίσουμε τα κενά και για να το πω πιο διανοικά ίσως τις αδυναμίες που υπογραμμίστηκαν και να κάνουμε τις απαραίτητες διορθώσεις. Να θυμίσω ότι είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε το θέμα της ε, ανθεκτικότητας, της αντίστασης στα αντιβιωτικά. Αυτό δεν ε, έχει να κάνει μόνο με τις διασυνοριακές απειλές, αλλά να δούμε ακριβώς την αντιμικροβιακή ε, ανθεκτικότητα και αντίσταση. Είναι μεγάλη μου, με μεγάλη μου ικανοποίηση, ακούω να συζητιέται ότι η πρόβλεψη κοινών αγορών είναι κάτι που μπορεί να λειτουργήσει για να οργανώσουμε καλύτερα μια κοινή αγορά. Αυτή η πλατφόρμα λοιπόν για την αγορά ε, συγκεκριμένων εμβολίων θα πρέπει να χρησιμοποιείται από τα κάτι μελη Μέχρι τώρα έχει κυρίως χρησιμοποιηθεί για την κοινή παροχή ιατρικού εξοπλισμού ε, και ιατροτεχνικών για την επιμέρους προστασία από μεταδοτικές ασθένειες για τους ασθενείς. Ακούω ότι είμαστε ήδη στο σωστό δρόμο. 14 κράτη-μέλη ήδη έχουν δεσμευτεί να συμμετάσχουν. Είναι τα μισά βέβαια από τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε αν θέλουμε να προχωρήσουμε κάπω πιο γρήγορα, θα ήταν καλό να ξέραμε τι ε, τρόπου χρησιμοποιούμε για να πείσουμε τα υπόλοιπα κράτη-μέλη να συμμετάσχουν και αυτά. Ευχαριστούμε. ο κύριο Πεντητσίνη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πρόλαβα. Η ανάγκη συντονισμένη αντίδραση για την υγειονομική ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αφορά μόνο τι πιο προφανεί απειλέ από τι μεταδοτικέ ασθένειε όπω η ΟΖΙΚΑ η έμπολα. Αλλά υπάρχουν και άλλα ζητήματα όπω η μικροβιακή αντοχή που είπε στην συνάδελφο. Εδώ λοιπόν χρειάζεται για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά όχι μόνο παρακολούθηση και ένα σύστημα ελέγχου που να είναι κατάλληλα και σκόπιμα, αλλά και συντονισμό μεταξύ των δράσεων και των αποκρίσεων στα μέτρα που χρειάζεται για να αναχαιτήσουμε αυτέ τι περιπτώσει. Μίλησα για την μικροβιακή αντοχή, αλλά όλο ιδιαίτερω θέλω να αναφερθώ τα αντιβιωτικά που χρησιμοποιούνται για τα ζώα και, που και τα, τα οποία ζώα προορίζονται για την ανθρώπινη κατανάλωση, την παραγωγή τροφίμων. Δηλαδή υπάρχει η σαλμονέλα, για να δώσω ένα απλό παράδειγμα, που μπορεί να είναι ανθεκτικά και να αντιστέκονται στα, μικρό, στα αντιβιωτικά και αυτές ε, οι μικροβιακές αιστείες να μεταδίδονται και στον άνθρωπο μέσω των τροφίμων. Εδώ λοιπόν κάτι πρέπει να προβλέψει η Ευρωπαϊκή Ένωση με ένα πρόγραμμα δράσης που να αναχαιτίζει να μας επιτρέπει να προστατευόμαστε από τις μεταδοτικέ ασθένειες με επίσημους ελέγχους, οι οποίοι να πραγματοποιούνται στα, σημεία ελέγχου των συνόρων. Επίσης, μια άλλη καταπήγουσα ανάγκη για τη δημόσια υγεία είναι η ε, πτώση της μικροβιακής προστασίας ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της μαζικής αύξησης μεταναστών. Δεν γίνεται να γίνει μαζικός για ασθένειες που στην Ευρώπη δεν απαντώνται τόσο πολύ όπως η πατήτιδα Α και Β, η φυματίωση, η ερυθρά, η διφθερίτιδα και άλλες ασθένειες. Οι μετανάστες θα πρέπει να εμβολιαστούν αμελητή με, προβλή, με προγράμματα εμβολιασμού ε, των εθνικών κρατών, όπως συζητήθηκαν την περασμένη εβδομάδα, όμως μπορεί και να διαφεύγουν από τα προγράμματα αυτά. Οπότε εκεί ε, μπορεί να υπάρχουν ε, προβλήματα λόγω των μεγάλων μεταναστευτικών ροών. Θα πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε συνολικά τι συμβαίνει. Πώς σκέφτεστε να επιλύσετε το πρόβλημα αυτό με μέτρα της δημόσιας υγείας, εφόσον ε, τέτοια αρμοδιότητα έχουν μόνο τα κράτη-μέλη. Και σε επίπεδο εθνικών κρατών μελών υπάρχει και κατακαιρματισμό επειδή τα μέτρα αυτά ε, προβλέπονται σε περιφερειακό επίπεδο. Ευχαριστούμε κυρία Τορνανό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η έκθεση αυτή θυμίζει σωστά ότι τα μέτρα δημόσιας υγείας που προβλέπονται για να αντιδράσουμε σε διασυνοριακές, σοβαρές διασυνοριακές απειλές και κινδύνους είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Το ίδιο και η, ολένα και μεγαλύτερη συμμετοχή των χωρών που είναι υποψήφιες για προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό πραγματικά με εκπλήσει. Είτε ως προς το να συμμετάσχουν στους ίδιους κανόνες, είτε στι διάφορε δοκιμέ για τη συγκέντρωση πληροφοριών και την σχετική πλατφόρμα για τη συλλογή δεδομένων για τις μεταδοτικές ασθένειες. Ήθελα λοιπόν να εμείνω στην σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων για την υγεία στο, στο, στα πλαίσια του συστήματο πρόορη ε, και έγκαιρη προειδοποίηση και αντίδραση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έκθεσή τη ε, αποφέρεται ότι η υπηρεσία στην έκθεσή τη πρέπει να εξασφαλίζει την αντικειμενικότητα των δεδομένων. Έτσι είναι, διότι ό,τι και να γίνει θα πρέπει να εφαρμοστούν οι ε, διεθνεί κανόνε υγεία. Αυτό είναι βέβαια μια αξιέπαινη πρόθεση, αλλά να μην ξεχνάμε ότι ο ίδιο ο ΠΟΗ ε, την περασμένη χρονιά, πέρσι, μα επέκρινε για την γραφειοκρατική διαχείριση της περσινής κρίσης. Ελπίζουμε λοιπόν ότι η ευρωπαϊκή αντίδραση στο συγκεκριμένο θέμα, παρά τις καλές προθέσεις που τη συνοδεύουν, θα μας οδηγήσει στο ίδιο αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Uh, εμείς ευχαριστούμε. Αν δεν θέλει άλλος κανείς το λόγο, να δώσω και πάλι το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Ράιν, για τις απαντήσεις. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις και τα σχόλιά σας. Θα ήθελα να επανέλθω σε μερικά σημεία. Καταρχήν, ω προ τι αδυναμίε και τα προβλήματα που εντοπίσαμε στην ετοιμότητα και πώ θα τα αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα και τι αδυναμίε. Στη σελίδα 5 τη έκθεση, εκεί σα παραπέμπω, προτείνουμε να επενδύσουμε από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Υγεία ε, σε κοινέ δράσει. Ένα καλό παράδειγμα θα ήταν ένα σχέδιο, ένα project για τη... τα υγειονομικά μέτρα στα πλοία που είναι ένα στενέ σημείο στις μεταδοτικέ ε, ασθένειε. Δηλαδή όλες οι λιμενικέ αρχέ των κρατών μελών μαζί με τις πλειοκτήτριε εταιρείε, είτε πρόκειται για επιβατικά πλοία είτε για εμπορικά, να δούμε πώ θα, βελτιώσουμε την, τον εντοπισμό και την ε, πρόληψη των μεταδοτικών ασθενειών, ιδιαίτερα στις θαλάσσιες μεταφορές. Εκεί εντοπίσαμε κάποιες αδυναμίες στο σύστημα ελέγχου και εκεί θα πρέπει να επενδύσουμε σε τέτοια προγράμματα. Επίσης ε, θα προβούμε σε αξιολογήσεις αναχώρα, γιατί άλλο να κάνει η ίδια χώρα μια αξιολόγηση για το πώς εφάρμοσε μια νομοθεσία και άλλο ένα ε, τρίτο εξωτερικό παρατηρητή να κάνει την αξιολόγηση. Εδώ υπάρχει ένα επιπλέον στοιχείο πίεση. Αυτή είναι μια δεύτερη πρωτοβουλία που σκοπεύουμε να αναλάβουμε. Δηλαδή να φέρουμε εξωτερικούς αξιολογητές για να ελέγξουν πώ λειτουργούν τα εργαστήρια και τι ικανότητε έχουν τα κράτη-μέλη να ανταποκριθούν. Αυτά είναι δύο παραδείγματα αλλά στη σελίδα 5 έχουμε και άλλα παραδείγματα πρωτοβουλειών που θα αναλάβουμε για να βελτιώσουμε την ετοιμότητα των κρατών μελών. Σε ό,τι αφορά τη μικροβιακή αντοχή που αναφέρθηκε δύο φορέ, αυτό είναι παγκόσμιο θέμα. Δεν επηρεάζει μόνο τη δημόσια υγεία, αλλά και την υγεία των ζώων, τη φαρμακοβιομηχανία, την έρευνα, την ερευνητική κοινότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θεσπίσει εδώ και χρόνια ένα σχέδιο δράση. Μάλιστα βρισκόμαστε στη φάση αξιολόγησης αυτού του σχεδίου δράσης για να προτείνουμε επιπλέον ή ε, ε, ενισχυμένα μέτρα για να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον τη μικροβιακή εντοχή. Και μάλιστα αργότερα μέσα στο έτος θα κάνουμε και κάποιες αναγγελίες σχετικά. Είναι σίγουρα ύψη προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η καταπολέμηση τη μικροβιακή αντοχής, γιατί είναι ουσιώδη ζήτημα ασφάλεια υγεία και όχι μόνο υγεία των ζώων, γιατί η χρήση των αντιβιωτικών στην κτηνοτροφία ε, επηρεάζει και την ανθρώπινη υγεία και εκεί είναι το πρόβλημα. Οπότε η προσέγγιση της ενιαίας υγείας, One Health Approach, είναι πάρα πολύ σημαντική και θα προτείνουμε πολλά μέτρα σχετικά. Επίσης έχουμε στενή συνεργασία με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας γιατί όσα μέτρα και αν έχουμε και όσο καλή και αν είμαστε στην Ευρώπη για τη μικροβιακή αντοχή, δεν θα μας ωφελήσει τίποτα αν όλο, όλος ο υπόλοιπος κόσμος υστερεί. Γι' αυτό μας ενδιαφέρει στενή συνεργασία και με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη μικροβιακή αντοχή και με τον Καναδά επίσης και με την Νορβηγία. Θέλουμε ε, χώρες ε, ισχυρή εταιρεία από την παγκόσμια κοινότητα να στηρίξουν τις προσπάθειές μας για την πάταξη της μικροβιακής ε, αντοχής. Αναφέρθηκαν ε, διφθερίτιδα, υπατήτιδα και κάποιες άλλες αρρώστιες που μπορεί να πλήξουν τους μετανάστες. Ε, ξεσπάσματα εξάρσεις τέτοιων μεταδοτικών νόσων σε πληθυσμούς προσφύγων που έχουν καταφέρει στην Ευρώπη του τελευταίους μήνες δεν οδήγησαν σε κατάσταση κρίσης. Ήταν μεμονωμένα παραδείγματα, απομονωμένα κρούσματα μεταδοτικών νόσων. Ο αριθμός των τραυματισμών αντίθετα εξαιτίας των συνθήκων διάπλου της Μεσογείου αυτό είναι πολύ πιο συχνό πρόβλημα από ότι οι μεταδοτικές νόσοι. Έχουμε και το επιπλέον πρόβλημα του άγχους ε, ή διαταραχές ε, εξαιτία του άγχους ε, από αυτό το επικίνδυνο ταξίδι που κάνουν του διάπλου της Μεσογείου. Πάντως ενισχύουμε το σύστημα ελέγχου, αλλά δεν είχαμε ανακοίνωση ιδιαίτερων κρουσμάτων μεταδοτικών ασθενειών από τους πρόσφυγες. Πάντως έχουμε ένα σύστημα ε, προαιρετικών μητρών υγείας, ώστε να επιτρέψουμε τους πρόσφυγες όταν ελέγχονται και καταγράφονται ε, να μπορούμε να κρατούμε ένα ιστορικό ε, της υγείας τους και όταν φτάσουν στο τελικό προορισμό τους να έχουν ήδη το προσωπικό τους ιατρικό μητρό. Αυτό εφαρμόζεται δοκιμαστικά στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή και θέλουμε να επεκτείνουμε αυτή τη χρήση του προαιρετικού μητρώου υγείας για τους πρόσφυγες, ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή μεταφορά από το σημείο άφηξη στο σημείο τελικού προορισμού, σε συνεργασία με την υπατερμοστή για τους πρόσφυγες, τα κράτη-μέλη και την ΠΟΕ. Τώρα, για την έγκαιρη προειδοποίηση, έχουμε έναν εξάρτητο οργανισμό που προστατεύει τα δεδομένα και κάναμε πολλές αλλαγές στο σύστημα για να το θωρακίσουμε θέλουμε και θωράκιση σε ό,τι αφορά την τεχνολογία των πληροφοριών, αλλά και τον έλεγχο των δικαιούχων της πρόσβασης στο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και αντίδρασης. Σε ό,τι αφορά την αντίδραση της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για τον έμπολα, τον ιό έμπολα, είχαμε μια έκθεση για τη Γενική Συνέλευση του ΠΟΗ σε ό,τι αφορά την αντίδραση του ΠΟΗ στην ε, επιδημία του έμπολα. Και επίσης ε, εξετάζουμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τις παγκόσμιες διατάξεις για την υγεία. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, προσπαθούν να βοηθήσουν την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας να βρει τρόπους για να, για να εφαρμόσει καλύτερα τις παγκόσμιες νομοθετικές διατάξεις για την υγεία. Και μάλιστα οι κυβερνήσεις από όλο τον κόσμο θα λάβουν μέρος τον επόμενο μήνα σε μια διάσκεψη της, Γενικής, ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ε, Γαλλικής Κυβέρνησης, ε, μια συνδιοργάνωση, ως συνεισφορά μας για να βοηθήσουμε την παγκόσμια κοινότητα να προβαίνει σε καλύτερη αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. Σας ευχαριστώ. Τώρα έχουμε ένα κενό. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα μέχρι τις 5 γιατί τότε περιμένουμε τον Αντιπρόεδρο Κατάινεν στις 5 η ώρα. Οπότε έχουμε 10-12 λεπτά. Ραντεβού εντός ολίγου. Dear colleagues, we have uh, suspended our meeting some minutes before. Συνάδελφοι, διακόψαμε πριν από λίγα λεπτά. Τώρα όμως είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι να ξαναρχίσουμε την συνεδρίασή μας. Καλωσορίζω θέμα τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Κατάινεν, εκ μέρου τη Επιτροπή ΕΝΒΗ. Ελπίζω να έχουμε μια υποφελή συζήτηση στα πλαίσια του επίσημου διαρθωμένου διαλόγου μα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ανυπομονώ να ακούσω για την υλοποίηση του προγράμματο εργασία σα για το 2016 και τι προτεραιότητέ σα πέραν τη χρονιά αυτή. Επίση, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι ο στόχο αυτή τη ανταλλαγή απόψεων είναι να μάθουμε τι γίνεται και με το πρόγραμμα δράσης για την οικονομία και την ε, υλοποίησή του. Ακόμα και πριν από αυτό το πρόγραμμα είχαμε, αποφασίσει να παρακολουθούμε στενά την εφαρμογή του. Γι' αυτό λοιπόν σας ευχαριστώ για την προθυμία σας να έρθετε και να ενημερώσετε την Επιτροπή μας για την πρόοδο που έχετε ε, καταφέρει να επιτύχετε και αυτό να γίνεται ένα εξάμενο. Σας ευχαριστώ για τη σημερινή σας παρουσία και σας δίνω πίσω μέσα στο λόγο. Για την ε, εισαγωγική σας παρέμβαση και μετά θα έχουμε τη συζήτηση με τους συναδέλφους τη Επιτροπής. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι βουλευτές, σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας και να ακούσω τις απόψει τη Επιτροπής ΕΝΒΗ για διάφορα ζητήματα. Ε, Όπω ξέρετε, η συνεργασία μα είναι πολύ στενή και η ε, Επιτροπή χαίρεται ιδιαίτερω να έχει διαρθρωμένο διάλογο με το Κοινοβούλιο. Μα ε, βοηθά αυτό να διαμορφώσουμε σωστά τι αποφάσει μα και να φωτίσουμε με ένα διαφορετικό τρόπο τις προτάσεις μας. Η δημόσια υγεία, το περιβάλλον και η προστασία των καταναλωτών είναι ένα θέμα που αφορά όλες μας τις πολιτικές και ένας τρόπος να πετύχουμε τους στόχους μας στην ατζέντα για την βιώσιμη ανάπτυξη για το 2030. Όμως, εκτός από τις μεταφορές και τη δημόσια υγεία, να ε, επικεντρωθώ τώρα σε δράσεις μας οριζόντιας φύσης, όπως την κυκλική οικονομία, το επενδυτικό πρόγραμμα και το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Πρώτα, δύο λόγια για τους ε, στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, που είναι το ευρύτερο πλαίσιο των δράσεών μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να έχει ηγετικό ρόλο στην ε, υλοποίηση και την παρακολούθηση τη ατζέντα για το 2030 τη βιώσιμη ανάπτυξη και το ίδιο και για του στόχου αυτή. Ανακοινώσαμε λοιπόν στο πρόγραμμα εργασιών μα για φέτο μια πρωτοβουλία για τα επόμενα βήματα που θα πρέπει να αντιληφθούν για το βιώσιμο ευρωπαϊκό μέλλον. Με την υλοποίηση τη ατζέντα των στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη στα πλαίσια τη αναθεώρηση ε, το 2020. Για να δούμε το κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο για τη βιωσιμότητα όλος ιδιαίτερος στις εσωτερικές μας πολιτικές ε, ως Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε αποφασίσει να επιδιώξουμε όλους τους στόχους ε, και σκοπούς ε, της, του θεματολογίου. Διότι συγκλίνουν και με του στόχου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ατζέντα του 2020. Τον έχουμε θέσει σε εργασία και απασχόληση για του Ευρωπαίου πολίτε και να βελτιώσουμε την αγωνιστικότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σαφή στόχο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και θα μα βοηθήσει να προχωρήσουμε ως Ευρώπη. Σε ό,τι αφορά την βιοποικιλότητα, επικεντρωνόμαστε στην ε, σαφή και με μικρότερο κόστος υλοποίηση του υπάρχοντος πλαισίου. Η ευρωπαϊκή βιωσιμότητα είναι μια ανάγκη προκειμένου να αντιμετωπίσουμε εθελοντικά μεγάλες προκλήσεις όπως την αποδυνάμωση των φυσικών πόρων και τη μεγαλύτερη συγκέντρωση των παρόχων ε, πόρων, τις δημογραφικές εξελίξεις και τις μετατοπίσεις δυνάμεων σε διεθνές επίπεδο. Για να λάβουμε αυτές τις προκλήσεις υπόψη θα πρέπει να δούμε τι συμβαίνει και από τη σκοπιά της ε, ε, σύγχρονης οικονομίας. Γι' αυτό και την οικονομία με ένα θεματολόγιο που θα μας επιτρέψει να δημιουργήσουμε περισσότερες θέσεις εργασία και να αντιμετωπίσουμε τις σχετικές προκλήσεις. Για την ίδια την πρωτοβουλία θα έχουμε μια λεπτομερή αξιολόγηση για να δούμε αν υπάρχουν κενά και λήψεις προς την επίτευξη των στόχων μας, όπως έχουν ανακοινωθεί στο θεματολόγιο του 2030. Αυτό θα είναι η βάση των συζητήσεών μα αργότερα φέτο. Μια συζήτηση που θα μα επιτρέψει να αποφασίσουμε τα επόμενα βήματα. Στο εντωμεταξύ θα συνεχίσουν οι αποφάσεις μας και θα υλοποιήσουμε επενδύσεις. Όπως το πακέτο της κυκλικής οικονομίας θέλουμε να μεταφραστεί σε πραγματικότητα και να προχωρήσουμε περισσότερο στην ενεργειακή αγορά. Ε, ενεργειακή στην εξωτερική διάσταση. Θα προσπαθήσουμε να βεβαιωθούμε ότι θα πετύχουμε το στόχο τη ατζέντα ε, του 2030 για την Ευρώπη και θα συνεργαστούμε μαζί σα για να γίνει αυτό επιτυχία. Στην κυκλική οικονομία τώρα. Μετά την παρουσίαση του πρώτου αντιπροέδρου Τίμερμαν και μου του ιδίου για το σχετικό πακέτο στην ε, ολομέλεια του Κοινοβουλίου στις 2 Δεκεμβρίου και την παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Επιτροπή στις 21 Δεκεμβρίου, με μεγάλη χαρά μπορώ να πω ότι οι συζητήσει στο Ευρωκοινοβούλιο έχουν προχωρήσει. Έχουν επικεντρωθεί και στο πρόγραμμα δράση και στι ε, συγκεκριμένε επιμέρου προτάσει μα. Είναι ενθαρρυντικό ότι θεωρείται τι προτάσει μα ω ένα ε, ολοκληρωμένο θεματολόγιο με σωστέ προτεραιότητε. Έχουμε 10 προτεραιότητε για την ώρα στα πλαίσια τη ευρύτερη, του ευρύτερου θεματολογίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τη δουλειά και την ανάπτυξη. Ε, το ίδιο στην ενέργεια και τις κλιματικές αλλαγές και εφόσον υπάρχει διεθνή συνένεση και δεσμεύσει για τι κλιματικέ αλλαγέ από το Παρίσι. Και ευρύτερα στο πλαίσιο θεματολογίου του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπω αποφασίστηκε και από τον ΟΗΕ το Σεπτέμβριο τη περσινή χρονιά. Η κυκλική οικονομία μπορεί να είναι μια πολύ μεγάλη συνεισφορά προ του δύο στόχου. Το πακέτο σχεδιάστηκε με βιώσιμε ευκαιρίε για τι επιχειρήσει. Αυτό ήταν το κέντρο των ενδιαφέροντό μα. Και επίση θελήσαμε να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των επιχειρήσεών τη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ήδη διεθνή πρωταγωνιστή στι πράσινε τεχνολογίε και λύσει και αν υπήρχε περισσότερο εξορθολογισμένη διαχείριση των πόρων, θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε την αποδυνάμωσή του και την ε, δική μα των τιμών σε διεθνή επίπεδο για να ενισχύσουμε ακριβώ την, το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα. Η καινοτομία είναι καθοριστική σημασία για την ανάπτυξη τη αγορά και να δημιουργηθούν θέσει απασχόληση και ε, ανάπτυξη, αλλά και να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητά μα. Πρέπει να κάνουμε κάθε προσπάθεια για να έχουμε υψηλέ επιδόσει στην ε, κατασκευαστικό τομέα που πρέπει να παραμείνει στην Ευρώπη με το σωστό πλαίσιο για τι επενδύσει, την καινοτομία και τι νέε τεχνολογίε καθώς και τις νέες τεχνολογικές λύσεις, οι οποίες θα μας επιτρέψουν να διαχειριστούμε την, ε, τους πόρους με εξορθολογημένο τρόπο βάσει των αρχών της κυκλικής οικονομίας, με ένα πλαίσιο φιλικό προς το χρήστη, τις ευρωπαϊκές εταιρείες και ιδίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα της κυκλικής οικονομίας θα πρέπει επίσης να παίξουν εδώ έναν ολοένα αυξανόμενο ρόλο. Με το Horizon 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επενδύει προ 600 650 εκατομμύρια ευρώ ε, για τους σκοπούς της κυκλικής οικονομίας. Πέραν αυτών, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει μια δέσμευση τριών δις ευρώ για την έρευνα και την κοινοτομία για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, των περιβάλλον, την ε, επαρκή χρήση των πόρων και τις πρώτες ύλες από το 2014 έως το 2020. Επιπλέον, ε, επικεντρωνόμαστε και στην υγεία αλλά και τι βιώσιμες εγκαταστάσεις και επενδύσει που θα πρέπει να διαφανούν στα πλαίσια του Στρατηγικού Ταμείου Επενδύσεων όπως και μέσα από τα διευθυντικά ταμεία. Ακόμη δοκιμάζουμε την ιδέα του να ξεκινήσουμε μια πλατφόρμα με τη συμμετοχή της Επενδυτικής, Ευρωπαϊκής Επενδυτικής Τράπεζας και των Εθνικών Τραπεζών για να ευνοηθούν οι στόχοι της κυκλικής οικονομίας. Υπάρχουν σημαντικές ε, σχέσεις συνεργασίας μεταξύ των βασικών νομοθετικών προτάσεων και του προγραμματος δράσης μας. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι αυτοί θα ενισχυθούν στη διαδικασία της συναπόφασης και ότι η υλοποίηση του προγράμματος δράσης θα προχωρήσει. Στο Συμβούλιο με πρωτοβουλία τη Ολλανδική Προεδρία, το πρόγραμμα δράση συζητήθηκε και σε περιβαλλοντικό επίπεδο, αλλά και από τη σκοπιά τη ανταγωνιστικότητα και στα ανάλογα συμβούλια, σε αυτού του σχηματισμού του Συμβουλίου. Καλωσορίζουμε τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στην όλη διαδικασία. Είναι σημαντικό να ακουστούν και δικέ σα απόψει για να συνεχιστεί η συνεργασία μα σε όλου του τομεί, προκειμένου να πετύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για όλα τα θεματολόγια που προανέφερα. Η δουλειά μα για την εφαρμογή του προγράμματο δράση έχει ξεκινήσει κάποια μέτρα πρόκειται να εγκριθούν ήδη φέτος. Ε, λόγου χάρη, η πρόταση για την αναθεώρηση των κανονισμών θα πρέπει να έρθει μάλλον την επόμενη, ε, τις επόμενες, για τα λοιπάσματα θα φτάσει τις επόμενες μέρες. Ε, πρέπει να έχουμε το κατάλληλο πλαίσιο για τι επενδύσει προκειμένου να εξασφαλίσουμε και τα απαραίτητα χρηματοδοτικά μέσα. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αποτελεσματικά το γενικότερο χρηματοδοτικό σύστημα ώστε να καλύψει του στόχου τη βιώσιμη ανάπτυξη και να πετύχουμε τι δεσμεύσει που αναλάβαμε πέρσι στη Σύνοδο Κορυφή των Παρισίων αλλά και στα πλαίσια του θεματολογίου του 2030 και του προγράμματος δράσης για την ευρωπαϊκή οικονομία. Η, αγορά, η Ένωση Κεφαλαίου Αγορών ε, περιλαμβάνει τη σαφή δεσμεύση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προωθήσει και να αυξήσει τη χρηματοδότηση για τους περιβαλλοντικούς και βιώσιμους στόχους και τις επενδύσεις τους. Θα συνεχίσουμε να εξετάζουμε το θέμα αυτό στη συνέχεια της χρονιάς σε συνάντηση που ονομάζεται «Επενδύοντας για ένα πρασινότερο μέλλον». Στο ΕΦΣΙ έχουμε εντοπίσει τι επενδύσει για την ε, προστασία των πόρων ω μια από τι βασικέ προτεραιότητε μαζί με την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Θα πρέπει να ε, ε, προωθηθούν τα περιβαλλοντικού, περιβαλλοντικού χαρακτήρα προγράμματα με στόχο να έχουμε μια πιο φιλική προς το περιβάλλον και με χαμηλότερη κατανάλωση άνθρακα οικονομία. Δύο παραδείγματα που θα χρηματοδοτηθούν από την ε, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι ένα πρόγραμμα στη Γαλλία για την οικοδόμηση και τη συνεργασία και άλλων ευρωπαϊκών αρχών με μία μονάδα για την ανακύκλωση και την κάψη αποβλήτων ε, ακόμη και επίσης για την αεροναυπηγική καθώς και την διασυνοριακή υδροδότηση ή τα προγράμματα ε, επεξεργασίας αποβλήτων μεταξύ περισσότερων των μία χωρών. Επίση, θα έχουμε σημαντικέ ευκαιρίε για τα μέλη και τι εταιρείε του μέσα από το ΕΦΣΥ, καθώ και για άλλου φορεί. Σε αυτό το πλαίσιο ε, είμαι πεπισμένο ότι πρέπει να μην φυστούμε καμία προσπάθεια για να προωθήσουμε την κοινοτομία και στον τομέα του περιβάλλοντο και τη δημόσια υγεία. Οι επιχειρηματίε γνωρίζουν ότι η προσοχή που δείχνουν ε, για το περιβάλλον του φέρνει περισσότερη δουλειά και έτσι θα μπορέσουν να αναπτύξουν τι επιχειρήσει του βιώσιμα και μακροπρόθεσμα. Αυτή τη στιγμή οι ευρωπαϊκέ εταιρείε δίνουν το 1 τρίτο των ε, πράσινων τεχνολογικών λύσεων σε διεθνέ επίπεδο. Και αυτό ελπίζουμε να πεντασπλασιαστεί το 2020. Η αγορά αυτή ολοένα μεγαλώνει και πρέπει να δράξουμε την ευκαιρία Ιδίω εφόσον στηρίξουμε τι επιχειρήσει μέσα από σαφεί πολιτικέ διαδικασίε που θα καθοδηγήσουν τι επενδύσει και θα τονώσουν την καινοτομία. Η πρόσφατη αναθεώρηση του οικολογικού προγράμματος του προγράμματος της οικολογικής δείχνει ότι η καινοτομία μπορεί να ενσωματωθεί στις περιβαλλοντικές πολιτικές. Η πράσινη λοιπόν καινοτομία πρέπει να συμπεριληφθεί ως διάσταση και σε υπόλοιπες, στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές πολιτικές. Υπάρχει και ένα σχετικό πρόγραμμα δράσης που δίνει, σημαντική, δίνει μεγάλη έμφαση ε, στην περαιτέρω ανάπτυξη της οικολογικής καινοτομία με την ευαισθητοποίηση, τη δημιουργία δικτύων, τη διαδικτύωση δηλαδή και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Αλλά και μεγαλύτερε χρηματοδοτικέ ευκαιρίε από του βασικού ενδιαφερομένου, τι μικρομεσαίε επιχειρήσει και τι αρχέ τοπική αποδίκηση των μέλων. Τα ίδια και για την υγεία. Η υγεία είναι ένα τομέα με μεγάλο δυναμικό για την ε, αναπροσέλκυση επενδύσεων και προκειμένου να εργαστούμε προ όφελο των πολιτών και των εταιριών. Δηλαδή υγεία για να υπάρξει και περισσότερη οικονομική ανάπτυξη και θέσει εργασία. Πρέπει να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να, ε, να επιδιώξουν τέτοιου στόχου για τις μικρομεσαίε τους επιχειρήσει. Η ηλεκτρονική επίση υγεία είναι που θα ενισχυθούν εφόσον υπάρξει την κατάλληλη μεταρρύθμιση των υγειονομικών συστημάτων. Ένα παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων επενδύει 70 εκατομμύρια ευρώ στην οικοδόμηση 14 νέων ε, κάποιων πρώτων κέντρων ε, στην Ιρλανδία, το οποίο θα έχει συνολικό κόστος 140 εκατομμύρια, αλλά χρηματοδοτήθηκε εν μέρει από τα και θα είναι μια, ένα από τα πρώτα μας προγράμματα. Ε, να επανέλθω σε μια άλλη οριζόντια προσπάθεια, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο είναι ένα σημαντικό όχημα για την περιβαλλοντική μας ε, ολοκλήρωση. Αλλά και τα υγειονομικά συστήματα μπορεί ε, να έχουν μεγαλύτερη βιωσιμότητα ε, και συνολική καθολική παροχή υπηρεσιών μαζί με την αλληλεγγύη που θα πρέπει να εκφραστεί ε, το 2016 πρέπει τα κράτη-μέλη να, λάβουν ε, δράση, να λάβουν δράση για την κυκλική οικονομία. Σε 18 από τις 26 αναχώρα ε, εκθέσεις που δημοσιεύτηκαν για την πρόοδο των κατομελών ως προς τους στόχους της οικονομίας και την εξορθολογισμένη διαχείριση των πόρων είναι στοιχεία που λάβαμε υπόψη. Επίσης στο πλαίσιο του εξαμήνου συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη για την αποτίμηση των υγειονομικών του συστημάτων και των αποδόσεων του ω προ την πρόσβαση, την αντεκτικότητα, την ποσότητα και την ε, βιωσιμότητα. Η πρόοδο αυτή θα επιτρέψει τα κράτη-μέλη να χαράξουν πιο τεκμηρωμένα την πολιτική του με τι κατάλληλε μεταρρυθμίσει εκεί που χρειάζονται. Ελπίζω ότι τα κράτη-μέλη θα μπορέσουν να μελετήσουν αυτέ τι προτεραιότητε στα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων, τα οποία περιμένουμε να δούμε τον Απρίλιο. Να ολοκληρώσω λέγοντα ότι έχουμε πολλέ ευκαιρίε να στηρίξουμε τη δημιουργία τη απασχόληση με νέε περιβαλλοντικέ ε, φιλικές πρωτοπεριβάλλον περιβάλλον και βιώσιμες λύσεις και πρέπει αυτό το δυναμικό να το εκμεταλλευτούμε πλήρως. Ευχαριστώ πολύ. Ε, σας ευχαριστούμε Αντιπρόεδρε Κατάινεν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίασή σας και τώρα να ξεκινήσουμε με τον πρώτο γύρο ερωταπαντήσεων με τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων. Να ζητήσω από τους συναδέλφους να είναι παρακαλώ σύντομοι και να δώσω πάρα αυτά το λόγο το κύριο Φλόρεντς από το ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Χάρηκα που αναφέρατε ότι ελπίζετε ότι τα κράτη-μέλη θα διακρίνουν τις ευκαιρίες που κρύβει η κυκλική οικονομία για αυτά και θα ήθελα να επενθυμίσω το εξής. Στην Ηνωμένα Έθνη αποφασίσαμε πρόσφατα για ένα πρόγραμμα εργασία σε το οποίο και αναφέρατε. Νομίζω λοιπόν ότι η Ευρώπη πραγματικά είναι σε καλό δρόμο στην ηγεσία. Και τώρα να αναφέρω και ποιε είναι οι ανησυχίε μου. Η κυκλική οικονομία είχε καταρρεύσει πριν από κάποια χρόνια. Δεν φταίγατε εσείς, ε, άλλοι. Άλλοι το είχαν προκαλέσει Τώρα λοιπόν όμως ε, έχει επανέλθει. Δεν ε, θεωρώ όμως ότι τονίζεται επαρκώς η κυκλική, οικονομία. Ένα παράδειγμα. Έχουμε εδώ πολλές εκθέσεις ε, οι οποίες πάντα ε, έχουν και προηγούμενες εκθέσεις και τέσσερις εκθέσεις που έχουμε εδώ μπροστά μας είναι συνέχεια παλαιών εκθέσεων με τις οποίες ασχολήθηκα δυστυχώ ή ευτυχώ. και αν κοιτάξουμε από τις προηγούμενες εκθέσεις τι έχει εφαρμοστεί ήδη καταστροφική κατάσταση. Ε, από πού βρίσκεται λοιπόν το θάρρος να μας λέτε ότι τα κράτη-μέλη βρίσκονται πλέον στο σωστό δρόμο για να τα εφαρμόσουν όλα αυτά. Γιατί στην τελική ανάλυση μιλάμε για τις πρώτες των παιδιών και των ε, εγγονιών μας. Αυτό θα πρέπει να το ανταλαμβανόμαστε, να το συνειδητοποιούμε, ότι δεν τσακωνόμαστε για το 60-65% Το θέμα είναι το κατά πόσο θα αρχίσει να ισχύει η οδηγία το 2030, το 2035. όποιο δεν τυπώνει σε σκέψει. δεν έχει καταλάβει τι περιλαμβάνει η έκθεση. Δεν πρέπει λοιπόν να μαλώνουμε και να πολεμάμε τα συγκεκριμένα ποσοστά. Θα πρέπει να ταρακουνήσουμε τα κράτη-μέλη και να τους πούμε ότι το θέμα είναι το συνολικό υλικό πρώτων υλών. Όχι κάποια Βράχει πρόθεσμα στα. Σας καλώ και σας προσκαλώ να ταρακουνήσετε τα κράτη-μέλη και ιδιαίτερα τις μεγάλες ε, χώρες. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε έτσι με τις πρώτες ύλες. Πού, πού θα βγάλουν λοιπόν τις πρώτες ύλες οι μελλοντικές γενιές. Ευχαριστώ. Thank you very much. And now for the social... Σας ευχαριστώ από του Σοσιαλιστέ, ο κύριο Κρότα. Ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Κατάνιαν για την ευκαιρία που μας δίνετε να διεξαγάγουμε διάλογο. Είσαστε υποδειγματικός. Μήπως θα μπορούσατε να πείτε και δύο λόγια στον κύριο Τίμερμανς, να σα μιμηθεί, για να μιλήσουμε και μαζί του, εδώ στην Επιτροπή. Γιατί είναι αρμόδιο για θέματα βιώσιμότητα και μπορεί λοιπόν να ακολουθεί το εξαιρετικό παράδειγμά σας για την ανταλλαγή απόψεων μαζί μας. Σε ό,τι αφορά το θέμα της κυκλικής οικονομίας. Νομίζω ότι είναι καλή η βάση, αλλά θα ήθελα να πω και να πάρω το μπαλάκι ε, που μας πέταξε ο συνάδελφος Φλόρεντς. Εφαρμογή, εφαρμογή. Να κάτσουμε και να σκεφτούμε πώς θα μπορούσαν να δημιουργηθούν και συνεργασίες, εταιρικέ σχέσεις. Ε, μίλησα με τους stakeholders, εμπλεκόμενους φορείς κτλ. Και πάντα ακούω το εξή ότι πάντα υπάρχει διάθεση για συνεργασία, διασυνοριακή, αλλά χρειάζεται και μια πλατφόρμα που να μας επιτρέπει. Πώς θα το πετύχουμε αυτό, μέσω το Ιντερεγ, δεν ξέρω. Αλλά υπάρχει όμως μια πλατφόρμα, γιατί υπάρχουν πολύ καλά παραδείγματα για το πώς η νομοθεσία μπορεί να εφαρμοστεί με σωστό τρόπο και νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό θα προχωρήσουμε ένα μεγάλο κομμάτι του δρόμου. Κάτι άλλο που ήθελα να αναφέρω σε ό,τι αφορά τη σπατάλη των τροφίμων. Αν θέλουμε να συναρπάσουμε τον κόσμο για την κυκλική οικονομία, καλά θα κάνουμε να βάλουμε στο επίκεντρο και να τονίσουμε και τη σπατάλη τροφίμων και να κάνουμε και μελέτες αντικτύπου για το πώς μπορούμε να αποτρέψουμε να σπαταλώνται ε, τροφήματα, ε, τα τρόφιμα, τα οποία τα πετάμε στα σκοπίδια, είναι πραγματικά και θέμα ηθικής αν θέλετε. Εκατό δισεκατομμύρια τόνοι για τα πρότυπα και την ε, σύγκληση των προτύπων. Πώς μπορούμε να τα πετύχουμε αυτό. Στην προκειμένη περίπτωση ε, έχουμε τις τιμές του πετρελαίου που είναι πάρα πολύ χαμηλές, καταστροφικό αυτό. Αλλά όταν θέλουμε να κάνουμε ανακύκλωση θέλουμε και πρότυπα. Πώς μπορούμε στο μέλλον να το, να το διαμορφώσουμε αυτό και τα δευτερογενή προϊόντα. Και ένα θέμα που με ε, απασχολεί πάρα πολύ το θέμα της ρήπανσης των θαλασσών, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το πλαστικό. Έχουμε πιο πολύ πλαστικό στις θάλασσες μας από τη ψάρια. Στη ρήπανση λοιπόν των θαλασσών θα πρέπει να κοιτάξουμε τι θα κάνουμε με τις πλαστικές σακούλες, γιατί ξεβράζουν στις ακτές στη Βορείο Θάλασσα, στην επικρατειά μου. Έχουμε προγράμματα για το πώς ε, μπορούμε να βγάλουμε το πλαστικό από τη θάλασσα. Σας παρακαλώ λοιπόν ε, βοηθήστε μας, υποστηρίξτε μας για να αποτρέψουμε για να δούμε τι θα κάνουμε με τις πλαστικές σακούλες, γιατί τα άλλα θα τα φάμε εμείς είναι τα πλαστικά που πετάμε στις θάλασσες. Ευχαριστώ, η κυρία Γκέρλινγκ. Σας ευχαριστώ και ευχαριστούμε κύριε Κατάνιν για την εισαγωγή που ήταν ευρύτατη, όπως και η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως και η όλη η αντίληψη περί κυκλικής οικονομίας. Είναι από τις πιο πολύ συζητημένες έννοιες των τελευταίων καιρών η κυκλική οικονομία. Αλλά θα πρέπει να δούμε πώς έχει πραγματικότητα. Και είναι κρίμα ε, που στην πρόταση δεν επισημαίνεται αυτό που ανέφερε ο κύριος Γκρούτε, Γκρότη και θα ήθελα να πω και εγώ. Τι γίνεται με την αξία της αγοράς ανακύκλωσης και πώς θα ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια ανακύκλωσης. 650 εκατομμύρια είπατε θα επενδυθούν σε προγράμματα επίδειξης, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και μια οικονομική απόδοση και με ενδιαφέρει κυρίως ο καταναλωτής, γιατί πολλοί που έχουν δει βουνά ολόκληρα πλαστικών που έχουν συγκεντρωθεί και μάλιστα με κόστος ε, και από την τσέπη του τοπικού αλλά δεν ανακυκλώνονται γιατί δεν υπάρχει αγορά για τη διάθεση αυτών των ανακυκλωμένων προϊόντων. Επίσης, ε, ε, σωρία χαρτιού που συγκεντρώνεται, το γνωρίζουμε στην Ηνωμένο Βασίλειο. Βέβαια ο κύριος λέει τα απόβλητα είναι ε, λεφτά, είναι χρήμα. Αλλά από ό,τι βλέπουμε προς το παρόν τα απορρίμματα είναι απλώς παθητικό. Και δυστυχώς δεν υπάρχει τίποτα στην πρόταση σας που προτείνει διόρθωση ε, βράχη και μέσο πρόθεσμα. Γιατί δυστυχώς ο κόσμος αρχίζει και χάνει την εμπιστοσύνη του στην, στο δυναμικό ανάπτυξη αυτής της αγοράς και επαφιόμαστε στους πολίτες ε, που τους ζητούμε να αλλάξουν τις συνήθειές τους, αλλά αν ε, δεν υπάρχει κάποια επιβράβευση, αυτό κάποια ανταβιβή, κάποιο ορατό αποτέλεσμα, δεν θα συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια αλλαγή. Η κυρία Γιαταρμάκη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, έχω δύο σύντομες ερωτήσεις. Το πρόγραμμα δράσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής λέει ότι η ενίσχυση η προώθηση της κυκλικής οικονομίας και η συναφής πρόοδος ε, θα γίνει σε στενή συνεργασία με τον Οργανισμό Περιβάλλοντος και τα κράτη-μέλη. Με στόχο, από ό,τι κατάλαβα, ένα απλό και αποτελεσματικό πλαίσιο ελέγχου. Τι πρόοδος έχει γίνει μέχρι τώρα στον τομέα αυτό. Δεύτερη ερώτηση. Για την ανοιχτή αγορά, ο καθοριστικός παράγοντας για την επιλογή του καταναλωτή είναι η τιμή. Και σε ό,τι αφορά το, τη ζήτηση των πρώτων υλών, ας μην ξεχνούμε ότι οι τιμές πολλών αγαθών και υπηρεσιών δεν αντικατοπτρίζονται στην διαδικασία αυτή. Και αυτό έχει και περιβαλλοντικές συνέπειες. Πώς λοιπόν θα μεριμνήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να συμπεριληφθούν και στην πράξη οι περιβαλλοντικές συνέπειες της κυκλικής οικονομίας στην τιμή του προϊόντος και να έχουμε μεγαλύτερη προβολή και διαφάνεια των αλυσίδων αξιών και να είμαστε σίγουροι ότι λαμβάνουν υπόψη και τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο και τις περιβαλλοντικές πτυχές. Αυτές τις δύο ερωτήσεις μόνο έχω. Ευχαριστώ. Ο κύριος Έκχολτ. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και τον Αντιπρόεδρο Κατάινεν για την επισκόπηση που μας έκανε. Οφείλω πάντως να ομολογήσω ότι συμφωνώ με τους ε, συναδέλφους, παρά ήταν γενική αυτή η επισκόπηση. Έχουμε βέβαια ένα σχέδιο δράσης, αλλά θέλαμε, θα θέλαμε να συζητήσουμε τι γενέστε με αυτό το σχέδιο δράσης. Και αυτό που μας είπατε είναι ότι μόνο η πρόταση αναθεώρηση ε, για τον κανονισμό για τα λοιπάσματα αναμένεται να δημοσιευθεί στο εγγυσ Τα υπόλοιπα στοιχεία του σχεδίου δράσης φαίνεται να καθυστερούν. Παρόλο που επικρίνεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι είναι πολύ καλή στη δημοσίευση εγγράφων εργασίας, μελετών και σχεδιοδράσεις, αλλά όταν ερχόμαστε στη φάση της δράσης, όταν θέλουμε να εφαρμόσουμε εμπράκτο στο σχέδιο δράσης, εκεί δεν έχουμε και πολλά. Τι γίνεται με το σχέδιο εργασίας για το οικολογικό σχεδιασμό, το eco design. Μας είχατε υποσχεθεί, αλλά ακόμη το περιμένουμε. Επίσης, συγκεκριμένη δράση ε, με βάση τους στόχου του 2030 για τον περιορισμό των απορριμμάτων και των αποβλήτων στη θάλασσα. Πού είναι. Περιμέναμε συγκεκριμένες προτάσεις ε, για τα διάφορα στάδια του σχεδίου δράσης και ομολογώ ότι δεν άκουσα τίποτα συγκεκριμένο στην παρέμβασή σας. Και αυτή την άποψη το πιο σημαντικό για μένα είναι τι συμβαίνει με τον οικολογικό σχεδιασμό. Γιατί πολλές φήμες ακούμε ότι ίσως οι καθυστερήσεις οφείλονται και στην εκστρατεία για το Brexit. Θα πρέπει όμως να εξηγήσουμε στον κόσμο προς τι αυτή η καθυστέρηση, γιατί θα πρέπει να το γνωρίζει ο κόσμος που οφείλεται η χρονοτριβή και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να είναι ο στόχος της συζήτησής μας. Και μια πιο γενική ερώτηση. Αναφερθήκατε στο εξάμεινο. Μας απογοήτευσε το γεγονός ότι στις προτάσεις δεν υπήρχαν συγκεκριμένα στοιχεία για το πώς μια οικονομία που θα αξιοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους τη συμπεριλαμβάνεται στο εξάμεινο. Πώς η κατανάλωση των πόρων θα είναι ένας από τους δείκτες που θα εφαρμοστεί στο εξάμεινο. Θα, θα μας μπορούσατε να το αναπτύξετε λίγο πιο διεξοδικά αυτό το σημείο. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Πεντιτσίνη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να πω ότι δεχτήκαμε θετικά το πρόγραμμα για την οικονομία της Επιτροπής για να μην έχουμε τέτοια υπερεκμετάλλευση των πόρων προκειμένου να ενισχύεται η υπερκατανάλωση. Έτσι οδηγήθηκαμε στη σημερινή περιβαλλοντική υποβάθμιση και την ελληπή διαχείριση αποβλήτων. Αυτά δεν μπορούν να συνεχιστούν. Όμως, κατά την άποψή μας, το πρόγραμμα δράσης πέραν των μέτρων που περιέχονται και έχουν προταθεί ήδη από χρόνια από την Επιτροπή, είναι αδύναμο. Σε καμία περίπτωση πλήρε. Εάν θέλουμε πραγματικά να υπάρξει την κοινωνική οικονομία, πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένε δράσει με συγκεκριμένου στόχου. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλό να προβλέψει λεπτομερή μέτρα με χρονοδιάγραμμα για την ε, εφαρμογή του με δύο βασικού πυλώνε. Ε, Όλε οι βλαβερέ επιδοτήσει ε, που μπορεί να βλέπουν το περιβάλλον να καταργηθούν. μεταξύ των οποίων αυτέ για το ρητά καύσιμα ή την καύση. Το ίδιο για το σύνολο του συστήματος παραγωγής. Ο στόχος δεν είναι η περισσότερη παραγωγή, αλλά η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση των υλικών και των προϊόντων. Μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει μια πραγματική μετάβαση προς την κυκλική οικονομία. Η ερώτησή μου λοιπόν προς εσάς, Επίτροπε, είναι απλούστατη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να έχει μια τέτοια προσέγγιση ή απλώς θα γυρίζουμε γύρω-γύρω από το πρόβλημα χωρίς να καταλήξουμε πότε είναι η πραγματική χωρις να καταληξουμε ποτε σε μια πραγματικη λυση Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ζάλκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, ήθελα να ξέρω για την τεχνική οικονομία. Ποια είναι η γνώμη της Επιτροπής για αυτό που έχει συνηθιστεί να ονομάζεται διαμεσολάβηση δηλαδή με άλλους ζώντες οργανισμούς να διαχειριζόμαστε τα απόβλητα. Αυτού του είδους η μεθοδολογία χρησιμοποιείται στην Ιαπωνία, στο Κιώτο, στο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα τη χώρα. Έχει δημιουργηθεί ένα τέτοιο βακτηρίδιο που χρησιμοποιείται για τις πλαστικές ύλε. Και εντάσσει μια αρχή του γνωστού, του διάσημου χημικού Λαβουαζιέ. δεν είναι η πρώτη τέτοια ο πρώτος τέτοιος χημικός τύπος που ε, χρησιμοποιείται, οι Ιάπωνες με τη χρήση αυτού του συστήματος κατάφεραν να διαλύσουν την πολυεφιλένη. 25 τόνοι ε, στην Ευρώπη ε, δεν ανακυκλώνονται. Εάν χρησιμοποιούσαμε λοιπόν μια τέτοια μεθοδολογία θα μπορούσαμε να έχουμε και μια ρεαλιστική λύση και ο τομείς τη έρευνα και τη καινοτομίας που είναι τόσο προσφυλή στην Επιτροπή να συγκλίνουν. Για την επιτυχία λοιπόν της κυκλικής οικονομία θα πρέπει να αναπτυχθεί η έρευνα της δύο διαμεσολάβσεις όπως έχει ονομαστεί. Αλλά με πραγματική εφαρμογή. Ε, ευχαριστούμε λοιπόν να μας πείτε την άποψή σα για το συγκεκριμένο θέμα. Ευχαριστούμε. Και τώρα μετά τον πρώτο γύρο ερωτήσεων των εκπροσώπων των διαφορών πολιτικών ομάδων, λόγω των αντιπρόεδρων Για να απαντήσετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις. Αυτές ήταν πολύ καλές και εύστοχες. Και θα προσπαθήσω να τις ομαδοποιήσω τις απαντήσεις μου. Αλλά παράλληλα θα προσπαθήσω να είμαι και όσο ακριβές γίνεται. Για την κυκλική οικονομία καταρχάς. Χαίρομαι που η Επιτροπή σας ενδιαφέρεται για όλο τον κύκλο γιατί είναι σαφές το πολιτικό μήνυμα από όλες τις πολιτικές ομάδες, αλλά και προς τον έξω κόσμο, ότι η κυκλική οικονομία θα αποτελέσει την κατεξοχήν τάση τις επόμενες, τα επόμενα χρόνια στο παγκόσμιο προσκήνιο. Γιατί το τρέχον μοντέλο, όπως σα είπα, φτάνει στο τέλος του, για πολλούς λόγους. Ακόμα και αν ε, του πήρε χρόνο να φτάσει στο τέλος του. Δεν έχει νόημα να το μείνουμε σε αυτό. Πόσο μάλλον που σκοπός μας είναι να διατηρήσουμε το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο. Κοινωνικό μοντέλο τι σημαίνει ότι θα πρέπει να αυξήσουμε την προσθεσμένη αξία. Προστιθέμενη αξία προέρχεται από την καινοτομία, από την παραγωγικότητα, αλλά και από την αποδοτικότητα στη χρήση των πόρων. Σήμερα λοιπόν η Ευρώπη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ενέκρινε μία ανακοίνωση για τη Χαλιβουργία. Μεγάλο θέμα, όπως ξέρετε όλοι σας. Αν ε, συγκρίνουμε όμως το γεγονός ότι στη ΣΥΠΑ η Χαλιβουργία είναι πιο αποτελεσματική ως προς τη χρήση της ενέργειας από ό,τι στην Ευρώπη, αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους αντιμετωπίζουν προβλήματα οι επιχειρήσει μα. Ο βασικό λόγο φυσικά είναι η υπερπαραγωγή που υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο. Αλλά αν μπορεί κανεί να παράγει το ίδιο προϊόν πιο αποτελεσματικά χρησιμοποιώντας λιγότερους πόρους, λιγότερη ενέργεια, αυτό ασφαλώς δίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Και αυτό μας καταδεικνύει με σαφήνεια το τι συζητάμε. Φυσικά δεν είναι αυτό το σύνολο των προβλημάτων και το σύνολο των θεμάτων που έχουμε να κάνουμε και αντιμετωπίζουμε στην ενέργεια. Είναι ένα μόνο θέμα. κοιτώντα του χρηματοοικονομικού πόρου που έχουμε στην ε, διάθεσή μα και που έχουμε ήδη δαπανίσει στην ε, κυκλική οικονομία ορίζοντα 2020. 650 εκατομμύρια για τα επόμενα δύο έτη για φέτος και για το 2014. 3-4 δισεκατομμύρια από τα τροφιτικά ταμεία ειδικά αφιερωμένα για την καλύτερη επεξεργασία. Τώρα κοιτάμε πώς θα δαπανίσουμε τα κονδύλια των τροφιτικών ταμείων. Πώς χρησιμοποιούνται λοιπόν τα κονδύλια αυτά. Δαπανούνται με καινοτομικού τρόπους για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των λιμάτων, τα αίτια, τα βαθύτερα αίτια των λιμάτων ή πρόκειται για μια έναν εξυγχρονισμό των ε, γεών, των ε, χιτά. Ελπίζω να ισχύει το πρώτο, να κοιτάμε το πώς μπορούμε να αποτρέψουμε την, την ε, παραγωγή ελλημάτων και το ΕΦΣΙ αποτελεί ένα καλό τρόπο για τις νέες επενδύσεις. Αλλά πέρα από τα χρήματα, η ρυθμιστική δύναμη την οποία έχουμε στα χέρια μας έχει τη σημασία της. Για τη κυκλική οικονομία τα περιβαλλοντικά ωφέλη είναι προφανή. Αλλά οι δύο αυτές λέξεις πραγματικά έχουν το νόημά τους. Κυκλική οικονομία και η ρυθμιστική εξουσία μπορεί να το πετύχει αυτό. Μπορούμε να εξασφαλίσουμε και να διασφαλίσουμε ότι προκύπτει από κάπου και κέρδος. άλλο δεν υπάρχει οικονομία. Και ε, οι αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο μπορούν να αλλάξουν και την κατεύθυνση όχι 100% αλλά εν μέρη α, την κατεύθυνση και την προέλευση του κέρδους. Γι' αυτό λοιπόν το ρυθμιστικό σκέλος είναι ακόμα πιο σημαντικό από ότι τα χρήματα, παρά το γεγονός ασφαλώς ότι πάντα για επενδύσει χρειάζονται χρήματα, αλλά αν το ρυθμιστικό πλαίσιο είναι σωστό, οι επενδύσει αποδίδουν κέρδος. Κύριε Φλόρενς, είπατε ότι η κυκλική οικονομία δεν εφαρμόζονται σωστά στα κράτη-μέλη. Αυτό αληθεύει. Στέκει. Αλλά ακόμα λιγότερο κατανοούν τα κράτη-μέλη τι ευκαιρίε που κρύβονται πριν από την κυκλική οικονομία. Γι' αυτό λοιπόν είναι μεγάλη πρόκληση τη ευαισθητοποίηση. Το θέμα τη ε, σπατάλη τροφίμων, κύριε Γκρότε, το θέσατε. Το αντιμετωπίζουμε και είναι τμήμα του σχεδίου δράση για την κυκλική οικονομία. Αλλά μία από τι δυσκολίε είναι η εξή. Δεν έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία για τη σπατάλη των τροφίμων, γιατί προέρχεται από διάφορες πηγές. Μας τα εστιατόρια, στα νοικοκυριά, από τον τομέα της λιανικής, της χοντρικής. Το προηγούμενο καλοκαίρι πήγα στη Μάλτα. Φανταστική χώρα, αλλά γενικά έχουν το συνήθειο να βγάζουν πολύ φαγητό. Πιο πολύ από ό,τι μπορεί να φάει ο καθένας. Αναρωτιόμουν λοιπόν, μα τι θα κάνουμε, θα έπρεπε να κάνουμε κάτι με αυτό το φαινόμενο. Είναι πολλοί οι λόγοι για τους οποίους έχουμε μεγάλη σπατάλη τροφίμων. Καταρχάς λοιπόν θα πρέπει να βρούμε τις πηγές της σπατάλης και μετά να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. σκοπεύουμε να βάλουμε και να συγκεντρώσουμε μια ομάδα εμπλεκομένων φορέων για να κάνουμε ένα σχετικό διάλογο για το ζήτημα τη πατάλης των τροφίμων. Είναι μεγάλη πρόκληση, σύμφωνοι. Δεύτερο θέμα και σε ό,τι αφορά τα δευτερογενή, τις δευτερογενείς πρώτες ύλες. Πολλοί βουλευτέ έθεσαν και το θέμα του, πλαστικού του πλαστικού. Έχουμε μια ενιαία αγορά για το πετρέλαιο, έχουμε μια ενιαία αγορά για το πλαστικό, δεν έχουμε όμως ενιαία αγορά, κοινή αγορά για το χρησιμοποιημένο πλαστικό. Και αυτό είναι μυστικό ζήτημα, ξέρετε και αποτελεί τον πυρήνα της κυκλικής οικονομίας. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε τα χρησιμοποιημένα υλικά, οι χρησιμοποιημένες πρώτες ύλες έχουν το ίδιο δικαίωμα να κυκλοφορούν διασυνοριακά όπως και οι πρώτες ύλες. Και αυτό ε, είναι, αν θέλετε, ο πυρήνα, η καρδιά τη κυκλική οικονομία Δεν υπάρχει κυκλική οικονομία αν δεν μπορούν και τα χρησιμοποιημένα, τα δευτερογενή αυτά προϊόντα να περάσουν διασυνοριακά. Αυτό εν μέρει οφείλεται στο γεγονό ότι κατατάσσονται ω ε, απόβλητα. Και τα απόβλητα την χάνουν διαφορετική αντιμετώπιση και μεταχείριση από την πρώτε ύλε. Αυτό λοιπόν είναι μια μεγάλη πρόκληση στην δημιουργία μια ενιαία αγορά για το πλαστικό. Η κυρία Γιατεμάκη έθεσε το ερώτημα του πώς ε, θα παρακολουθήσουμε το σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία και την εφαρμογή του. Όταν θα καταθέσουμε τις προτάσεις μας και όταν οι συνομοθέτες ε, εγκρίνουν τις προτάσεις μας, θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε και το ευρωπαϊκό εξάμεινο ως ένα εργαλείο να παρακολουθήσουμε το πόσο και καλά εφαρμόζουν και πετυχαίνουν τους στόχους στα κράτη-μέλη. Ίσως το πιο απλό που θα μπορούσαμε να παρακολουθήσουμε θα ήταν η πρόταση για τα απόβλητα όταν θα εγκριθεί από τους νομοθετές. Είναι αρκετά εύκολο και απλό να παρακολουθήσουμε ποια θα είναι τα επόμενα βήματα που θα λάβουν τα κράτη-μέλη για να μειώσουν τον όγκο των αποβλήτων που καταλήγει σε χωματερές και τι γίνεται και με την ανακύκλωση. Αυτό λοιπόν ε, θα αποτελούσε μια λύση για τις τιμές των πρώτων υλών τώρα και για τις τιμές των προϊόντων. Είναι σημαντικές ασφαλώς όταν οι καταναλωτές επιλέγουν ε, τα προϊόντα που θέλουν να καταναλώσουν. Δεν είμαι βεβαίω αν μπορώ να απαντήσω στο ερώτημα που μα θέσατε επαρκώ, Αλλά και πάλι το ρυθμιστικό πλαίσιο είναι καθοριστικό στην προκειμένη περίπτωση, γιατί η τιμή των πρώτων υλών ακολουθεί το ρυθμιστικό πλαίσιο εν μέρη. Αν ε, θέσουμε πρότυπα για κάποια συγκεκριμένα για κάποιε συγκεκριμένε πρώτε ύλε. Για παράδειγμα, για το καδμίο, το επίπεδο καδμίου στην οδηγία για τα λοιπάσματα. Αν ε, μειώσουμε το επίπεδο λοιπόν πρακτικότητα του καδμίου και δώσουμε τη δυνατότητα στου αγρότες, στου καταναλωτέ, να επιλέξουν διαφορετικά προϊόντα, είναι ένα βήμα. Κύριε Eichhout, είπατε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καθυστερήσει σε ό,τι αφορά το σχέδιο δράση. Δεν είμαι σίγουρο ότι έχουμε καθυστερήσει, αλλά ξέρετε πάντα παίρνει χρόνο να προετοιμαστούν οι συγκεκριμένε προτάσει προ του συνομοθέτε. Εγκρίναμε το σχέδιο δράση στι αρχέ Δεκεμβρίου και έκτοτε. Προετοιμάζουμε λοιπόν το σχέδιο δράση. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα παράλληλα, γιατί έχουμε και περιορισμένο αριθμό υπαλλήλων στι διάφορε γενικέ διευθύνσει. Αλλά όπως σας είπα, οι πρώτες συγκεκριμένες προτάσεις θα αφορούν την οδηγία για τα λοιπάσματα, σε ό,τι αφορά δηλαδή την αναθεώρηση. σε ό,τι αφορά τη συνεκτική στρατηγική για το πλαστικό για το επόμενο έτος. Θα καλύψει το συνολικό κύκλο και όχι μόνο ένα τμήμα αυτό. για τα επόμενα δύο χρόνια για τον οικολογικό σχεδιασμό και το σχετικό σχέδιο δράση. Θα το ολοκληρώσουμε το συντομότερο δυνατόν. Δεν μπορώ να σα δώσω μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Το συντομότερο δυνατόν. Αυτό που είναι πιο σημαντικό όμω ε, για το σχέδιο δράση είναι το πώ μπορούμε να διαβρύνουμε... Ε, το πεδίο εφαρμογή τη σχετική οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα αλλαγέ στην νομοθεσία. Απλά θα πρέπει να αποφασίσουμε πώ θα λάβουμε υπόψη την αποδοτικότητα των πόρων, όχι μόνο την αποδοτικότητα στην κατανάλωση τη ενέργεια. Γιατί η οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό είναι πάρα πολύ σημαντική για να δώσει πραγματική εξουσία, δύναμη στον καταναλωτή. Από τη στιγμή που ο καταναλωτή θα ξεκινήσει να επιλέγει διάφορε υπηρεσίε παραγωγή, και νέα αγορά. Και θα ανακατευθυνθεί η πηγή του κέρδους σε ό,τι αφορά τις εταιρείες. Θα επανέλθουμε όμως το θέμα αυτό στο εγγύς μέλλον. Τώρα για τη νέα τεχνολογία με τη, βιολογική, τη χρήση βιολογικών οργανισμών. Δεν έχω γνώσει. Θα προτιμούσα να μελετήσω πρώτα το θέμα για να μην πω κάτι απροετοίμαστος. Πάντως φαίνεται καλή πρόταση, ενδιαφέρουσα να χρησιμοποιήσουμε την καινοτομία. Αλλά δυστυχώς δεν έχω αρκετές γνώσεις για να σχολιάσω. Τώρα, πώς μπορούμε να περιλάβουμε την κατανάλωση των προώρων στο ευρωπαϊκό εξάμεινο. Το έχω σκεφτεί, αλλά σίγουρα δεν είναι και το πιο εύκολο ζήτημα. Ε, ας πάρουμε για παράδειγμα μια χώρα που παράγει ξυλία για την παραγωγή χάρτου και χαρτοπολτού. Και άλλη χώρα καταναλώνει αυτό το χαρτί και το χαρτοπολτό. Σε ποιο ισολογισμό, σε ποιες χώρες στον ισολογισμό θα υπολογιστούν αυτοί οι πόροι. Αυτό είναι ένα απλό παράδειγμα. Αλλά αν δείτε την αλυσίδα αξιών, ε, διαπιστώνετε ότι μπορεί να είναι αρκετά εκτεταμένη. Οπότε, ποιο θα θεωρούμε ότι χρησιμοποιεί τους πόρους, αυτοί που τους, αυτός που τους, τους, παράγει, αυτός που τους καταναλώνει. Θα πρέπει να έχουμε σαφή βάση δεδομένων με δείκτες και μετά να αποφασίσουμε σε ποιο ισολογισμό, στο ισολογισμό ποιας χώρας θα προσυπολογιστεί η κατανάλωση των πόρων. Ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στο δεύτερο γύρο. Παρακαλώ συνάδελφοι να είστε λακωνικοί γιατί 15 ζητήσατε το λόγο και σε 3 τέταρτα πρέπει να ολοκληρώσουμε. Κύριε Γκροστέτ, ευχαριστώ Κύριε Επίτροπε, ακούγοντας σας, διαρωτόμαστε κατά πόσο λαμβάνετε υπόψη την πραγματικότητα. Όταν είπατε ότι θα ήταν πιο ανταγωνιστική αν ε, καταναλώναμε λιγότερη ενέργεια. Ε, στα χαλιβουργία για παράδειγμα. Επισκεφτόμαστε όμως τα χαλιβουργία και διαπιστώνουμε ότι ήδη οι χαλιβουργίες έκαναν τεράστιες προσπάθειες για να περιορίσουν την ε, κατανάλωση ενέργειας. Και παρόλα αυτά δεν καταφέρουν να είναι ανταγωνιστικές σε σχέση με τον εισαγόμενο χάλιβα. Οπότε υπάρχει δυσκολία. Παρά τις προσπάθειες δεν έχει αναβαθμιστεί η ανταγωνιστικότητα. Επίσης συναντήθηκα στην εκλογική μου περιφέρεια με μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ήδη έχουν ε, εμπλακεί σε αυτή την κυκλική οικονομία. Έχουν τεράστιο πρόβλημα όμως με τη διέξοδο, με τη διάθεση στην αγορά. Είναι έτοιμες να λάβουν δράσεις, να αναπτύξουν τις πρωτοβουλίες τους και τις δραστηριότητές τους στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας, αλλά χρειάζονται διέξοδο και μάλιστα σχετικά κοντά στον τόπο παραγωγής. Και αυτό είναι το πιο δύσκολο. Να έχουμε σωστή οργάνωση ώστε να δημιουργηθούν αγορές. Γιατί είναι αγαθές οι προθέσεις της κυκλικής οικονομίας και όλοι αισθενιζόμαστε αυτή τη βούληση για την κυκλική οικονομία. Αλλά υπάρχει με τεράστιο χάσμα μεταξύ θεωρίας και πράξης, προθέσεων και εφαρμογής. Αυτό θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε. Και τι εργαλεία έχουμε στη διάθεσή μας για να εξασφαλίσουμε τέτοιες διεξόδους, ώστε να υλοποιήσουμε αυτή την κυκλική οικονομία σε συγκεκριμένη περιφέρεια και έκταση. Η κυρία Μποναφέ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ που στην παρέμβασή σας αλλά και στις απαντήσεις σας Κάνατε πολλέ αναφορέ στι δυνατότητε τη κυκλική οικονομία, ένα ανταγωνιστικό φέλο για το πλεονέκτημα μάλλον για το οικονομικό μα σύστημα και την δυνατότητα να έχουμε νέε επενδύσει σε καινοτομία, σε τεχνολογικέ λύσει για να ανακάμψει η απασχόληση, η απασχόληση ποιότητα. Αυτέ τι παρατηρήσει σα τι συμμερίζομαι απολύτω. Όμω θα μου επιτρέψετε, μια και μιλάμε για την εφαρμογή του προγράμματο δράση, θα μου επιτρέψετε και θα με συγχωρήσετε να επιτρέψω σε ένα θέμα που εξετάστηκε κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Περιβάλλοντο και Ανταγωνιστικότητα και επειδή προέκυψαν κάποια ερωτήματα. Είναι μια καλή ευκαιρία για να επαναλάβω μια αρχή που θέλω να μα καθοδηγεί και να εξηγηθώ. Εάν θέλουμε πραγματικά να υπάρξει μετάβαση προ την κοινωνική οικονομία, το πρόγραμμα δράση είναι μια ιδρυτική, θα έλεγα, θεμελιώδη πράξη για να προχωρήσουμε. Ιδάλω θα πρέπει να αναθεωρηθούν τέσσερι οδηγίε για την χρήση, τη διαχείριση των αποβλήτων, αλλά αυτό είναι τελείω διαφορετικό δεν έχει να κάνει με την κυκλική οικονομία, γιατί δεν μιλάμε για κυκλική βιομηχανία έτσι κι Θέλουμε η κυκλική οικονομία να δώσει ένα νέο μοντέλο για ολόκληρη τη βιομηχανία και την παραγωγή τη στην Ευρώπη. Όμω το πρόγραμμα δράση έχει κεντρικό ρόλο η κυκλική οικονομία, αλλά το ίδιο θα έπρεπε να συμβαίνει και με, την, με τον οικολογικό σχεδιασμό. Δηλαδή πρόβλεψη του παραγωγή προϊόντων που να είναι συμβατά με του οικολογικού μα στόχου. Η κυκλική οικονομία δηλαδή πρέπει να κοιτάξει και τα προϊόντα στην προέλευσή του, τη δυνατότητα τα προϊόντα να επαναχρησιμοποιούνται και να ανακυκλώνονται. Όλα αυτά, τα είπατε κι εσεί, έχουν να κάνουν με την κοινοτομία. Την κοινοτομία στι επιχειρήσει, τα συστήματα, αλλά ε, μακροπρόθεσμα και όλου του στόχου που θέλουμε να πετύχουμε. Υπό το φω λοιπόν των όσων είπατε ότι θέλετε να επιδιώξετε, διαρωτώ με. Το είχαμε προτείνει και στο ψήφισμα Πιτικάινεν για την οδηγία με τον οικολογικό σχεδιασμό, eco-design, που για την ώρα αφορά μόνο τα ενεργειακά προϊόντα, αλλά θέλουμε να συμπεριλαμβάνονται όλα τα προϊόντα που έχουν σχέση με την κίνηση των πόρων. Στο πρόγραμμα δράση σα προτείνατε ε, εφαρμοστικέ πράξει. Όμω, εάν ε, σκεφτούμε τι μέσο πρέπει να χρησιμοποιηθεί, εσεί είπατε ότι χρειάζεται χρόνο. Για μένα δεν είναι ο χρόνο αυτό που λείπει. Ό,τι ε, χρειαστεί να γίνει πρέπει να γίνει άμεσα. Διότι πρέπει να καλύψουμε το κενό και να επικεντρωθούμε σε ένα συγκεκριμένο στόχο, αλλά ακριβώ δεν πρέπει να παραμένουμε μόνο στην ιδρυτική πράξη τη πολιτική οικονομία, αλλά και σε αυτήν του οικολογικού σχεδιασμού των προϊόντων. Ευχαριστούμε κυρία Βυσνιάσκα. Ευχαριστώ και κύριε Αντιπρόεδρε και κύριε Επίτροπε. Είναι αναμφίβολο ότι η ιδέα καλύτερης αξιοποίησης των πρώτων υλών και ελαχιστοποίηση των απορριμμάτων και των αποβλήτων στην καθημερινότητα είναι αγαθή πρόθεση και σωστή κατεύθυνση. Η ιδέα ε, της κυκλικής οικονομίας είναι πολύ σημαντική και μπορεί να είναι η κατάλληλη λύση. Σωστή κατεύθυνση και φαίνονται αρκετά φιλόδοξοι οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρά είναι όμως φιλόδοξοι για τις νέες χώρες. Ε, φαίνεται το, αντελήφθη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γι' αυτό και παρέτεινε κατά μία πενταετία τη μεταβατική για μερικές χώρες. Μερικές χώρες όμως με παρόμοιους δείκτες παραγωγής, ιδιαίτερα για τα ε, λίματα, όπως είναι η Τσεχία, η Πολωνία, η Ουγγαρία, η Βουλγαρία, δεν έχουν τέτοιες δυνατότητες. Και η Σλοβακία, η Ελλάδα ή η Λετωνία έχουν λάβει εξαιρέσεις. Ε, γιατί ε, δεν έγινε και για τις υπόλοιπες χώρες. Μήπως θα πρέπει να τύχει μεγαλύτερη διαφοροποίηση η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες των κρατών μελών, ιδιαίτερα για τα αστικά λύματα. Αναφέρεται το 2030 ε, και το δίκτυ το 65%. 64% ε, έχει η Γερμανία, 20% έχει η Πολωνία. Μέχρι το 2030 είναι δυνατό να καλύψουμε σχεδόν 45% και να φτάσουμε στο ίδιο αποτέλεσμα Γερμανία και Πολωνία ενώ ξεκινάμε από τόσο διαφορετικά ποσοστά. Θα χρειαζόταν μεγαλύτερη διαφοροποίηση πρότασή σας. Ευχαριστώ. Η κυρία Μέισνερ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και τον κύριο Επίτροπο. Μία παρατήρηση έχω να κάνω μετά από αυτά που είπε ο κύριο Ματία Γκρότ. όντω, στο μέλλον ε, θα χρειαστούμε πιο πολλά για την ε, ενέργεια για την διατροφή και για το καθεξής. Και αν δεν έχουμε ένα υγιεινό τρόπο, θα έχουμε προβλήματα. Λοιπόν, τρεις ερωτήσεις έχω να κάνω σε ό,τι αφορά την κυκλική οικονομία, κυρίως σε ό,τι αφορά τις πανίες Αυτό συμπεριλαμβάνεται στις προτάσεις σας για την κυκλική οικονομία, ότι η βιομηχανία θα πρέπει να παράγει προϊόντα τα οποία θα κρατούν πιο πολύ. Ναι, ρωτώ όμω, τι λέει η ίδια η βιομηχανία οικονομικό κράτο και πιστεύετε ότι σε ό,τι αφορά τι ε, σπανίε γέε θα αρκέσουν και δεν θα χρειαστεί να αρχίσουμε να ψάχνουμε στον πυθμένα της θάλασσης. Κατά δεύτερον, σε ό,τι αφορά το χαρτί ως ε, πρώτη ύλη. Από το ξύλο είναι πρώτη ύλη και συμβατική ύλη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την κατασκευή διάφορων προϊόντων. Τρίτη ερώτηση, η χαλιβουργία την αναφέρατε σε ό,τι αφορά την κυκλική οικονομία, ο χάλιβας είναι καλός γιατί μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά και ξανά. Αλλά είναι ε, υψηλής ε, κατανάλωσης ενέργειας. Πώς ε, πιστεύετε ότι θα εξελιχθεί η σημασία του χάλιβα λοιπόν στο μέλλον, δεδομένου ότι και στην Ευρώπη δεν είναι πολύ παραγωγική η παραγωγή, πολύ παραγωγή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λέω κύριε Σεμπαούντς. Δεν μπορώ να είμαι πεντάχο παρόν, γι' αυτό και έχασα ένα τμήμα της παρέμβασης. Θα ήθελα, κύριε Κατάινεν, να ζητήσω μεγαλύτερη φιλοδοξία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για την κυκλική οικονομία και για τη διαχείριση των αποβλήτων. Είπατε ότι είστε φιλόδοξοι. Πιστεύω ότι θα μπορούσατε να είστε ακόμη περισσότερο φιλόδοξοι. Από τις τελευταίες μας συνεδριάσεις διαπιστώνουμε με ανησυχία ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, υποβαθμίζει τα κριτήριά της και τις γενικές διατάξεις. Στην τελευταία ε, συνάντηση που είχαμε φάνηκε ότι μετριάστηκαν οι φιλοδοξίες για την αποτέφρωση για παράδειγμα. Θα σας θέλω παρακαλούσα μη χαλαρώνετε την ε, πίεση και τη φιλοδοξία. Βέβαια υπάρχουν και εθνικέ αρμοδιότητε, ναι. αλλά δεν θα πρέπει αυτέ να τροχοπεδίσουν τι φιλοδοξίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό ακριβώ θα πρέπει να είστε ακόμη πιο φιλόδοξοι στη, στη θέσπιση των στόχων και των προτεραιοτήτων. Όπω είπα, χρειαζόμαστε ένα πιο φιλόδοξο πακέτο μέτρων. Για παράδειγμα, για τη διαχείριση των αποβλήτων. Θέλουμε δεσμευτικού στόχου και βράχη και μέσο πρόθεσμα και να μην παρατείνουμε υπερβολικά τις προθεσμίες και τις μεταβατικές περιόδους. Μάλιστα υπάρχουν κάποια ευρωπαϊκά εδάφη που απέδειξαν την ικανότητα να ανταποκριθούν και χωρίς υψηλές φιλοδοξίες δεν πρόκειται να υλοποιήσουμε τη συστημική αλλαγή που τόσο χρειαζόμαστε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φλέκ. Ε, ε, κύριε Σκύρλετς, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο, τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που μας παρουσίασε το πακέτο για την κυκλική οικονομία και έχω δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις και ελπίζω ότι θα μου δώσετε και κατάλληλες και ικανοποιητικέ απαντήσεις. Η πρώτη ερώτηση αφορά αυτό που είπατε και στην ομιλία σας στην αρχική. Δηλαδή, ε, η λήψη υπόψη της ε, αποτελεσματικότητας των πόρων στο ευρωπαϊκό εξάμεινο. Η αποτελεσματικότητα, η αξιοποίηση, η αποτελεσματική χρήση των πόρων είναι πολύ σημαντικό θέμα και το επισήμαναν και τα Ηνωμένα Έθνη, αν και είναι απογοητευτικό ότι εμείς έχουμε μείνει πίσω σε σχέση με τα Ηνωμένα Έθνη. Πάντως, αν αφήσουμε κατά μέρο τα στοιχεία, ε, για να είμαστε αποτελεσματικοί και στο ευρωπαϊκό εξάμεινο πρέπει να έχουμε δείκτες της αποτελεσματικότητας. Για παράδειγμα θα μπορούσαμε να δούμε τα στατιστικά στοιχεία, αλλά εδώ έχουμε 28 διαφορετικές μεθόδους συγκέντρωσης στατιστικών δεδομένων που φτάνουν στη Eurostat. Οπότε και εσείς και εμείς με βάση αυτά τα στοιχεία λαμβάνουμε κάποιες αποφάσεις, κάνουμε κάποιες επιλογές και στην οικονομία. Αλλά δεν είναι ομοιόμορφη η μεθοδολογία συγκέντρωση αυτών των στατιστικών δεδομένων πρόκειται να αναλάβετε κάποιες πρωτοβουλίες για να εναρμονίσετε τις μεθοδολογίες ή να καταλήξετε σε μια ενιαία μεθοδολογία για τη συγκέντρωση αυτών των στατιστικών δεδομένων από τα κράτη-μέλη. Επίσης, ε, για, τα, για τις δευτερογενείς ύλες. Πρόβλημα, ένα πρόβλημα που υπάρχει είναι η διαφορά μεταξύ των εθνικών διατάξεων των κρατών μελών. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των, εθνικών, εθνικών νομοθεσιών. Σε μερικά κράτη τα απορρίμματα, τα απόβλητα θεωρούνται πόροι παρά σκουπίδια. Υπάρχουν όμως κανονιστικά προβλήματα με τη διάθεση στην αγορά και το κανονιστικό πρόβλημα δεν αφορά το ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά το εθνικό επίπεδο. Πώς θα ε, λυθούν αυτά τα προβλήματα, γιατί μπορεί να έχετε καλές προθέσεις, αλλά δεν αρκούν για να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα, το να μετατρέψουμε τα απόβλητα σε πόρους. Ευχαριστώ. Η κυρία Κέστιγκερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και εσάς, κύριε Επίτροπε για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση για ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα και νομίζω ότι σίγουρα θα λάβατε μεγάλη υποστήριξη από δική μας πλευρά γιατί πραγματικά, μόνο μια πραγματικά κυκλική οικονομία ε, θα μπορέσει να προωθήσει την αρχή της βιωσιοτιμότητας που φυσικά υποστηρίζουμε όλοι. Μία συγκεκριμένη ερώτηση έχω να κάνω σε ό,τι αφορά τα λήματα σε ό,τι αφορά τη συμπερίληψη του κριτηρίου της ποσότητας του όγκου που αναφέρεται. Αυτό τι θα σήμαινε για τα ξενοδοχεία και για τα εστιατόρια. Θα τα από την ε, διάταξη αυτή για ό,τι αφορά δηλαδή την ε, μεταφορά των αποβλήτων. Αυτό θα έπρεπε να γίνει από τους ιδιώτες και όχι από τους δήμους. Και αυτό θα σημαίνει αύξηση του κόστου. Δεν είμαι βέβαιη λοιπόν ότι θα ήταν σκόπιμο κάτι τέτοιο. Και μια και λειτουργεί καλά το σύστημα, γιατί δεν το αλλάξουμε. Μια δεύτερη ερώτηση σε ό,τι αφορά τον περιορισμό τη ποσότητα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια αιτιολόγηση. Τι είχατε κατά νου. Δεύτερη ερώτηση. Για τα βιολογικά απόβλητα. Σε ό,τι αφορά την ξεχωριστή συλλογή των βιολογικών αποβλήτων. Υπάρχει κάτι πολύ θετικό. Στην Αυστρία υπάρχει αυτή η αρχή για τη μείωση των αποβλήτων αυτών, αλλά δυστυχώς και τα πλαστικά σε πολλές περιπτώσεις συγκαταλέγονται στα βιολογικά και πάλι θα πρέπει να περάσουν από ε, από δεύτερο ξεχώρισμα. Είναι δηλαδή ουσιαστικά μόνο θεωρητικά βιολογικά πολιτά και στην πράξη πρέπει να ξεχωριστούν πριν γίνει η αποτέφρωση. Γι' αυτό λοιπόν εδώ θα ήθελα να σας ρωτήσω μήπως και εδώ υπάρχει κάποια λύση για να καταστεί πιο πρακτική αυτή η ρυθμίση. Όταν μιλάμε λοιπόν για την κυκλική οικονομία και όταν κοιτάμε το, τις σχετικές διατάξεις να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε στο βαθμό του δυνατού τη γραφειοκρατία. Αλλά σα ευχαριστώ πάρα πολύ σε κάθε περίπτωση και μπορείτε σίγουρα να υπολογίζετε στην υποστήριξη από πλευρά μα. Ευχαριστώ και τώρα ο κ. Λάινεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, Αντιπρόεδρε Κατά. Είναι ορίσατε και καλώς ορίζω μάλλον την έκκλησή σας να περάσει η έννοια της κυκλικής οικονομίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Την επόμενη εβδομάδα έχω προσκληθεί στην Κίνα για να μιλήσω για την κυκλική οικονομία. Η ερώτηση λοιπόν που έχω να απευθύνω είναι η εξή. Υπάρχει κάτι σε κλιματική διπλωματία. Υπάρχει κάτι αντίστοιχο σε ό,τι την κυκλική οικονομία, γιατί σε μία μέρα, κάποια μέρα θα χρειαστούμε και πρότυπα και προδιαγραφέ για τα ανακυκλωμένα σε ό,τι αφορά την κυκλική οικονομία. Δεύτερη ερώτηση. Κάποιοι συνάδελφοι το έθιξαν και αυτοί είναι ότι χρειαζόμαστε ιδιωτικέ επενδύσει. Πώ λοιπόν θα προωθήσουμε τι ιδιωτικέ επενδύσει, Νομίζω ότι χρειαζόμαστε και κίνητρα και ζητήματα τα οποία θα αποτρέψουν. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε και από πλευρά φορολογική πολιτική. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Ντεμάσμέικερ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, Επίτροπε, 1η Μαρτίου συμμετείχα σε μια συζήτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις λύσεις βάσει της φύσης, όπου και πάλι ζητήθηκε να κοιτάξουμε τι γίνεται και με τις πρώτες ύλες, γιατί στην παρούσα φάση χρησιμοποιούμε 1,5 φορές στον πλανήτη μας ε, και ζούμε και καταναλώνουμε μελλοντικέ ε, πηγές και μελλοντικέ πρώτες ύλες. και αυτό αποτελεί προτεραιότητα. Η καλύτερη κατανάλωση, η καλύτερη χρήση των ε, πρώτων υλών αποτελεί προϋπόθεση για την αγωνιστικότητα της Ευρώπης. Ό,τι και επιχειρήματα και να υπάρχουν όμως, η συγκεκριμένη δράση θα πρέπει να ακολουθήσει εκ των υστέρων. Και έτσι λοιπόν ερωτώ, πώς μπορείτε να συμβάλλετε προκειμένου να τονίσετε ακόμα πιο πολύ την ανταγωνιστικότητα με έργα και με πράξεις την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς μπορούμε να ε, δουλέψουμε εγκάυσια σε όλους τους τομείς της πολιτικής, προκειμένου μακροπρόθεσμα να προωθήσουμε αυτή την οικονομία και πώς μπορούμε να προωθήσουμε τις λύσεις ε, τις φυσικές. Και επίσης ε, να τονίσω κλείνοντας ότι όλα αυτά συνάδουν και με την ατζέντα για το 2030. Και ποια είναι τα βήματα που θα κάνετε βράχη πρόθεσμα για να εφαρμοστεί αυτή η ατζέντα για το 2030 και να συνδεθεί με την στρατηγική για το 2020 σε ό,τι αφορά την κυκλική οικονομία. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Γκζίμπ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ο Επίτροπος είπε ότι από τις πρώτες νομοθετικές πρωτοβουλίες για την κυκλική οικονομία θα είναι η οδηγία για τα λοιπάσματα. Ε, και η περιεκτικότητα καδμίου στα λοιπάσματα με φωσφορούχα, με άλατα. Από τις πληροφορίες που έχουμε λάβει από τον κλάδο, ε, φαίνεται ότι, φαίνεται ότι τα επίπεδα είναι αρκετά φιλόδοξα, αλλά μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πληρεί αυτές τις ε, υψηλές προδιαγραφές για τα φωσφορούχα άλατα και την περιεκτικότητα του καδμίου στα λοιπάσματα. Οπότε, τόσο φιλόδοξοι στόχοι που θα περιληφθούν στον κανονισμό για τα λοιπάσματα στα ρωσοφιλανδικά σύνορα είναι ρεαλιστικό να περιμένουμε να εφαρμοστούν. Μια και οι γειτονικέ χώρε δεν θα εφαρμόζουν αντίθετα κριτήρια. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα επίπεδα ανακύκλωση των πλαστικών. Πρόκειται για πολυμερές προϊόν, οπότε η ανακύκλωση μερικές φορές είναι αδύνατη και μερικές φορές από την ανακύκλωση γίνεται τοξικό. Οπότε λαμβάνετε υπόψη αυτό το στοιχείο των τοξικών πλαστικών τις απαιτήσει που έχετε για την ανακύκλωση και στις προτάσεις που θα υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τέλος. Για την διάρθρωση των αποβλήτων και των απορριμμάτων στα κράτη-μέλη. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές και στη διάρθρωση και στην περιεκτικότητα. Για παράδειγμα, στην Πολωνία 72% των αποβλήτων είναι βιομηχανικής προέλευσης από τον ενεργειακό κλάδο ή από τις εξορυκτικές βιομηχανίες. Αυτό είναι ένα μεγάλο ποσοστό των αποβλήτων. Οπότε είναι αξιέπαινοι οι φιλόδοξοι στόχοι, αλλά για παράδειγμα ο στόχος για την διάθεση των οργανικών αποβλήτων, για παράδειγμα. Δεν θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ε, και την πιθανότητα να φτάσουν και αυτοί ε, στα, στα ρεύματα, γιατί θα μπορούσαν και αυτά να χρησιμοποιηθούν για ανακύκλωση. Οπότε οι γενικές διατάξεις δεν θα πρέπει να έχουν αρνητικά αποτελέσματα και τα δύο απόβλητα που φτάνουν ε, στο, στη ροή των αποβλήτων ε, να είναι αδύνατον να αξιοποιηθούν στα πλαίσια μιας βιοοικονομίας. Ήταν κρίμα να τα χάσουμε αυτά τα βιολογικά απόβλητα. Επίσης θα πρέπει να διευκολύνουμε την τοπική αυτοδιοίκηση, τις τοπικούς και περιφερειακούς φορείς γιατί θα είναι δύσκολο με τόσο υψηλού στόχου οι τοπικοί και περιφερειακοί φορεί να καταφέρουν να σεβαστούν την κοινωνική νομοθεσία. Ευχαριστώ κυρία Σύρια Πέρικ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πρόεδρε ε, Πίτροπε, να σας πω ότι στη Ολλανδία είμαστε πάρα πολύ θετικοί για την ε, κυκλική οικονομία. Εξαιρετικά ε, ενθαρρυντικοί αλλά καθημερινά βλέπω επιχειρηματίε κόσμο που δεν ξέρουν προ τα πού πρέπει να πάνε, προς τα πού πρέπει να οδεύσουν. Νομίζω ότι χρειάζεται λοιπόν σωστή ενημέρωση. Το πρώτο θέμα. Χρόνια περιμέναμε λοιπόν την αναθεώρηση τη ε, οδηγία για τα λοιπάσματα από το 2003-2004 σε ό,τι αφορά ε, τα όλα, θέματα, όλα τα θέματα που μα απασχολούν. Αλλά χθε άκουσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν υπάρχει το θέμα της ε, μεταφορές από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Ε, τι πρέπει να κάνουμε για να το πετύχουμε αυτό. Πρόκειται για βιολογικά λοιπάσματα σε ό,τι αφορά τα λοιπάσματα στις θάλασσες τώρα. Από πλευρά της ε, Ολλανδίας, μία α, εταιρεία έχει πλοία τα οποία μαζεύουν τα πλαστικά στη θάλασσα. Όλα αυτά είναι θετικά. Τα γνωρίζετε λοιπόν όλα αυτά. Μιλήσατε επίσης συνάδελφε για την Κίνα. Εξ όσων κατάλαβα, στην Κίνα ο ΦΠΑ για την κυκλική οικονομία είναι με μηδενικό συντελεστή. Αυτό έχει μεγάλη διαφορά. Μπορούμε στην Ευρώπη να συμφωνήσουμε κάτι μεταξύ μας, γιατί και αυτό θα έχει θετικό αντίκτυπο. Και τέλος, μιλήσατε για τα τρόφιμα, για τη σπατάλη, για το μαγείρεμα. Το θέμα είναι πώς ε, οργανώνει κανείς τη διατροφή του στο σπίτι, στο νοικοκυριό. Δεν χρειάζεται να τα πετάει. Μπορεί να τρώει μία μέρα την εβδομάδα τα υπόλοιπα. Πολλά λοιπόν μπορούμε να συμφωνήσουμε και να πετύχουμε μαζί. Δεν χρειάζεται καν να μπουν όλα αυτά στην νομοθεσία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, λέει και ο Πρόεδρο. Η κυρία Ντελέη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω δύο θέματα, αλλά είναι πολύ συγκεκριμένα. Είμαστε στο μήνα Μάρτιο και τα μέτρα αυτά έχουν ανακοινωθεί για το 2016. Θέλω να ξέρω πώ έχετε προχωρήσει. Επίση, ε, μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα ήταν ε, λογικό να προβλέψετε έναν ιστότοπο ώστε οι πολίτες ε, που τους αφορούν τα θέματα αυτά να μπορούν να ενημερώνονται και να ξέρουν πώς προχωρείτε και να ξέρετε ποιε είναι οι κοινέ ε, πρόοδοι που επιτυγχάνεται. Η διάρθρωση των νέων και υπερχόντων μέτρων θα είναι σημαντική. Όπως ε, για την σήμανση των ε, οικολογικών και περιβαλλοντικών διαστάσεων υπάρχουν ήδη σήματα οικολογικά και περιβαλλοντικά. Μην δημιουργήσουμε νέα πρότυπα, πρότυπα που να μην ταιριάζουν με αυτά που ήδη υπάρχουν και ένα πιο συγκεκριμένο θέμα που έθιξαν οι συνάδελφοι, η καταπολέμηση της διασπάθησης τροφίμων. Ε, χρειάζεται εδώ ένα σαφή και συγκεκριμένο ορισμό. Δεν μπορούμε να αγωνιστούμε αποτελεσματικά και δραστικά ή να ε, καταμετρήσουμε την πρόοδο. Μπορείτε να μα πείτε πώ θέλετε να προχωρήσει για την εφαρμογή μια κοινή μεθοδολογία εφόσον αναφέρετε και το θέμα των ροών και τη αξιολόγηση του όγκου, ε, νομίζω ε, ότι σημαντικό είναι να υπάρξει ένα ορισμό ε, συγκεκριμένο στη διασπάθηση την υπερκατανάλωση τροφίμων. Ένα απλό παράδειγμα. Μήλα. Ένα μήλο που, που ε, έχει ξαπίσει είναι κατάλληλο για κατανάλωση γιατί έχει μικροτοξίνες. Δύο λοιπόν επιλογές. Ή θα προτείνεται από θρεπτική σκοπιά, από τη σκοπιά της διατροφής έναν ορισμό, οπότε σε αυτή την περίπτωση ήταν απόβλητο, αλλά ε, εάν ο ορισμός είναι ευρύτερος, το μήλο αυτό δεν μπορεί να καταναλωθεί από τον άνθρωπο, όμως μπορεί παρόλα να χρησιμοποιηθεί ως βιομάζα, οπότε να παράγει αέριο. Σε αυτή την περίπτωση δεν είναι πλέον απόβλητο, ούτε θεωρείται ότι σπαταλά, ε, σπαταλάτε. Οπότε, σπαταλείται Αυτό μου φαίνεται πολύ σημαντικό λοιπόν ω προ τον ορισμό των αποβλήτων. Επίση, βλέπουμε σε πολλά κράτη-μέλη όπω τη Γαλλία, την Ιταλία και την Δανία. Γίνεται μεγάλη μελέτη για αυτό το θέμα τη διασπάθηση και σπατάληση τροφίμων. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε τι καλέ πρακτικέ των διαφορών κρατών μελών με τη συμμετοχή και των ενδιαφερομένων φορέων. Τέλο, Νομίζω ότι πέρα των πρωτοβουλίων που λαμβάνουν τα κατημέλη, η Ευρώπη έχει έναν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει. Πρώτον, μπορούμε να επιδιώξουμε του στόχου βιώσιμη ανάπτυξη από κοινού για τον το χρονικό ορίζοντα του 2030. Έπειτα να ενερμονίσουμε του ευρωπαϊκού κανόνε και εκεί ε, σκέφτομαι όλο ιδιαίτερα το θέμα του νερού και των τροφίμων. Και ακόμη ε, νωρίτερα θα έλεγα ότι το θέμα είναι η ιεράρχηση των αποβλήτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και μία παρατήρηση για να ολοκληρώσω. Θα έλεγα ότι είναι κάπως γενικότερη ε, και για να επιστήσω την προσοχή των συναδέλφων και για την ε, σωστή εξέταση του θέματος νομίζω σκόπιμο θα ήταν να έχετε μια συμβολή λίγο πιο συγκεκριμένη και μάλιστα γραπτή με συγκεκριμένες προτάσεις για το τι ακριβώς θα κάνετε στο πρόγραμμα εργασιών σας ε, και να ενημερωθούν έτσι όλοι οι βουλευτές. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρος. Και τώρα ολοκληρώσαμε τον κατάλογο των μιλητών και θα δώσουμε το λόγο στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής για να λάβουμε και κάποιες απαντήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε διάφορες ερωτήσεις και διάφορα σχόλια για τα οποία ουσιαστικά δεν μπορώ να δώσω απαντήσεις, αν και μπορώ να υποκριθώ ότι κάτι απαντώ. Αν χρειάζεται επιπλέον διευκρινήσεις ευχαρίστως να σας τις δώσουμε εγγράφους. Και να ξεκινήσω με την παρατηρήση της κ. Κρουστέτ ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή χαλιβουργία, ότι είναι ενεργειακά αποδοτική. Αυτό στέκει. Πολλές εταιρείες ε, έχουν περιορίσει την κατανάλωση ενέργειας και γενικώ ε, σε γενικέ γραμμέ ισχύει αυτό. Τα πάμε καλά. Αλλά φυσικά υπάρχουν και εταιρείε που δεν είναι πολύ αποδοτικέ σε ό,τι αφορά την κατανάλωση ενέργειας και υπάρχουν και μεγάλε διαφορέ μεταξύ των χωρών. Και αν προσθεθεί και η διάσταση της διαφοράς ε, της τιμής της ενέργειας στα διάφορα κράτη-μέλη, γιατί υπάρχουν και μεγάλοι συντελεστέ φορολόγηση σε κάποιες χώρες και αυτό σημαίνει ότι ο ηλεκτρισμός είναι πολύ ακριβώς και αυτό δημιουργεί φυσικά επιπτώσεις για την ανταγωνιστικότητα. Το βασικό όμως θέμα σε ό,τι αφορά το χάλιβα είναι ότι στην Κίνα, λόγω της Κίνας, έχουμε υπερπαραγωγή διπλάσια σε σχέση με την συνολική παραγωγή της Ευρώπης. Αυτό είναι το θέμα με, τα, τον χάλβα από την Κίνα. Σε ό,τι αφορά την κύκλικη οικονομία, για όσους ενδιαφέρονται για το θέμα αυτό, να πω ότι εγκρίναμε μια ανακοίνωση σε ό,τι αφορά τα εμπορικά ζητήματα, τα εμπορικά μέτρα και τα εμπορικά εργαλεία. Θα τα διαβιβάσουμε και στα κρατημέλη. για να εγκρίνει το Συμβούλιο την, ε, τον εξυγχρονισμό των ε, μέσων ε, προστασίας του εμπορίου. Πώς μπορούμε να δώσουμε τώρα διόδους και διάβλους για τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με την κυκλική, με την κυκλική οικονομία. Δεν ξέρω αν μπορεί να το κάνει αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά τη δημιουργία διάβλων προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να ευαισθητοποιηθεί εν μέρη ο καταναλωτής για την ε, βιώσιμη παραγωγή στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας και αυτό που μπορούμε να κάνουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να χρησιμοποιήσουμε τις ρυθμιστικές εξουσίες σε ό,τι αφορά την επισήμανση, για παράδειγμα, της ενέργειας. Θα μπορούσε να υπάρχει πιο ευρύ εφαρμογή στον οικολογικό σχεδιασμό. Όταν ο καταναλωτή ξεκινά και επιλέγει διάφορα προϊόντα, δημιουργεί αυτό μια νέα πηγή κέρδου και αυτό αλλάζει την αγορά. Έτσι πάνε τα πράγματα. Ε, επισκεφτήκα στη Σουηδία νεαρούς επιχειρηματίες που παράγουν ε, ρούχα. Ρούχα πάρα πολύ μοντέρνα από ανακυκλωμένες ύλες. Μπορούν λοιπόν τα ρούχα όταν έχουν χαλάσει αν θέλετε να επιστραφούν στα μαγαζιά για να ξαναχρησιμοποιηθούν. Υπάρχει μια τέτοια ανακύκλωση και μάλιστα αυτό είναι πολύ στη μόδα, ξέρετε, στη Σουηδία. Εμείς ως πολιτικοί πάντα έχουμε την τάση να θέλουμε να επιλύσουμε όλα τα προβλήματα, αλλά θα πρέπει να είμαστε και ταπεινόφρονες και να αναγνωρίζουμε ότι δεν μπορούμε να λύνουμε όλα τα προβλήματα, απλά να, να δημιουργούμε το σωστό περιβάλλον στο οποίο ο κόσμος θα μπορεί να λαμβάνει τις αποφάσεις του ανάλογα και με τα μέσα που έχει στη διάθεσή του. Γι' αυτό λοιπόν η οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό είναι και τόσο σημαντική και για τις μικρομεσαίες εκείνες που θέλουν να παράγουν από δευτερογενείς ύλες. Ιδιαίτερα με το πλαστικό έχουμε πρόβλημα, όπως είπατε, το οποίο δεν μπορεί να περάσει τα σύνορα γιατί θεωρείται ως θεωρείται αποβλητό. Η κυκλική οικονομία επίσης ε, είναι και θέμα ασφαλώς εσωτερικής αγοράς. Πώς μπορούν οι χώρες τώρα να βελτιώσουν την διαχείριση των αποβλήτων και των λιμάτων. Υπάρχουν δεσμευτικοί στόχοι. Ελπίζουμε να το αποτεχθούν αυτό οι συνομοθέτε. και έχουμε και έναν διάμεσο στόχο που έχουμε θέσει. Οι χώρες εκείνε που υστερούν που δεν μπορούν να κινηθούν όσο γρήγορα θα έπρεπε. Για τις χώρες λοιπόν αυτές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ζητήσει να καταθέσουν ένα σχέδιο για το πώς θα πετύχουν τους στόχους εγκαίρως. Και αυτό μας βοηθά να βοηθήσουμε τα κρατημέλη να χρησιμοποιήσουν τις βέλτιστες πρακτικές, να τις διαδώσουμε τις βέλτιστες πρακτικές από τις άλλες χώρες. για το πώς μπορούμε να πετύχουμε τους ειδικούς στόχους. Αν καταφέρουμε λοιπόν να αποφασίσουμε για το πακέτο για τα απόβλητα των συντομότερο δυνατόν, θεωρώ ότι η Ευρώπη θα βρεθεί σε εντελώ διαφορετική κατάσταση σε σχέση με τη σημερινή σε ό,τι αφορά την ανακύκλωση και σε ό,τι αφορά τα απόβλητα που πηγαίνουν στους χωματερές. Σε πολλές περιπτώσεις ακούω και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο όταν συζητώνται διάφορα ζητήματα πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι. Δεν θέλω να γίνω γενής. Απλώς να πω ότι γίνομαι κάπως, αρχίζω να γίνομαι αλλεργικός σε αυτήν την ε, έκφραση. Πιο φιλόδοξος. Ε, πάντα καλό είναι να είναι κανείς πιο φιλόδοξος, αλλά θέλω να επιστήσω την προσοχή στην υλοποίηση. Αυτό είναι το θέμα. Πρέπει να είμαστε πραγματιστές για να πετύχουμε αποτελέσματα το θεματολόγιο του τουρκικού νομίζω όπω το προτείναμε είναι μια καλή αρχή. Δεν αλλάζει τον κόσμο διαμιά. Είναι σημαντικό ότι έχουμε όμω μια καλή αρχή, έχουμε μια δομή προσπαθώντα να καλύψουμε όλο τον κύκλο. Ε, θα ήθελα να έχουμε κάποια πρώτα αποτελέσματα. Η οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό, πώ να την αξιοποιήσουμε καλύτερα από ό,τι κάνουμε τώρα. Θέλω να δω αποτελέσματα για του στόχου για τι χωματερέ, τα αρχήτα. Ε, για την διεθνή των αποβλήτων. Θέλω να δω πόσο γρήγορα μπορούμε να προχωρήσουμε και να έχουμε μια νέα αγορά αποβλήτων για το πλαστικό και ούτω καθεξής. Δηλαδή ας επικεντρωθούμε λιγάκι στα αποτελέσματα και αν δούμε ότι κάτι πετυχαίνουμε τότε ανεβάζουμε τον πύχη, τον ανεβάζουμε ετησίω. Αλλά δεν μπορεί το θεματολόγιο της κυκλικής οικονομίας να τα κάνει όλα από την αρχή. Είναι σίγουρα πολύ ε, έχει πολλά στοιχεία, ε, δεν είναι όμω πλήρε και α επικεντρωθούμε στα πρώτα αποτελέσματα. Καταλαβαίνω ότι θέλετε να είμαστε πιο φιλόδοξοι, αλλά α πρώτα τα εφαρμόσουμε και μετά κοιτάζουμε τη φιλοδοξία. this resource efficiency target database and methodology. Ως προς τους στόχους, τη βάση δεδομένων και τη μεθοδολογία μας. Συζητάμε με τη Eurostat πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη βάση δεδομένων, τι ζητάμε από τα κράτη-μέλη και ποιοι είναι οι σωστοί δείκτες που πρέπει να χρησιμοποιούνται. Αυτά όλα είναι βασικά θέματα. Οι δείκτες ε, αφορούν τις βασικές εγκαταστάσεις. Ε, είναι τα θεμέλια μας αν θέλουμε να βελτιώσουμε τη διαχείριση των πόρων. Θέλουμε με την ψηφιακή οικονομία. Πρέπει να υπάρχει πρόσβαση στην ευρυζωνικότητα. Πρέπει να ξέρουμε πόσους πόρους καταναλώνουμε, πόσους χρησιμοποιούμε. Αυτά κάνουμε και επιδιώκουμε στη συνεργασία μας με τη Eurostat. Ε, στα αποβλήτα και τη διαχείριση αποβλήτων συνήθως, εάν κατάλαβα ε, καλά, μιλήσατε για τις χωματερές ε, ταχύτητα δημοτικές από που τα διαχειρίζονται δημοτικές αρχές ή τέλο πάντων σε περιφερειακό επίπεδο. Θα υπολογίζονται και αυτά μαζί με τα απόβλητα των Δήμων, όμω οι επιχειρήσει όπω οι τουριστικέ θα πρέπει να προσαρμοστούν στο νέο περιβάλλον των αποβλήτων και των απορριμμάτων. Πρέπει να αλλάξουν τι πρακτικέ του. Πρέπει να μειώσουν τα απόβλητα και αν υπάρχουν να τα ανακυκλώνουν όσο μπορούν. Κόστος θα υπάρξει. Αλλά τα πάντα εξαρτώνται και από την ιδεοντολογία τη κάθε επιχείρηση. Για την ε, διεθνή διάσταση, πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Δεν ξέρω και δεν έχω πληροφορηθεί ακόμα για αυτό που λέτε, αλλά στην Κίνα υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσε μελέτε. Έχουν κάποιο είδου στόχου ε, στο πενταετέ του πρόγραμμα και την περασμένη φορά που επισκέφτηκα τη χώρα συζητήσαμε για τι επενδύσει και την κυκλική οικονομία και θέλω να ακούσουν τι κάνει η Ευρώπη αλλά θα έλεγα ότι μάλλον εμεί πρέπει να κοιτάξουμε το τι κάνουν εκείνοι. Καταλαβαίνω από αυτό που σχολιάσατε βέβαια ότι με το πρόθεσμα θέλουμε περισσότερο εναρμονισμένη συνολική ε, κατάρτιση προτύπων έστω ή έστω ηθική ε, την προσέγγιση μα, δηλαδή τη φιλοσοφία μα προ το θέμα. Για τι επενδύσει, τι είδου επενδύσει, ρυθμιστικέ αλλαγέ δίνουν καλύτερα κίνητρα από ό,τι λόγω χάρη τα φορολογικά μέτρα. Τα φορολογικά μέτρα πάντοτε δυσκολεύουν το, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν θέλουμε να αλλάξουμε ε, τους κανονισμούς μας, πρέπει να αλλάξει και το επιχειρηματικό μας μοντέλο. Το θέμα των λοιπασμάτων. Η πρότασή μας παραμένει ανοιχτή. Θα προτείνουμε να μειωθούν τα επίπεδα καθμίου διότι θέλουμε να υπάρχει ίσως ανταγωνισμός μεταξύ των ε, από ανανεώσιμες πηγές ή ανακυκλωμένα λιπάσματα και των ε, λιπασμάτων και των συμβατικών. Δεν ξέρω αν είναι πολύ φιλοδοξός ο στόχος μας, όμως η πρότασή μας θα είναι ένας συνδυασμός, μια συμβαστική λύση των διαφορών απόψεων που υπάρχουν στην Επιτροπή και μεταξύ των δύο συνομοθετών. Ο στόχος είναι να δημιουργήσουν μια νέα αγορά για τα οικολογικά λιπάσματα. Υπάρχουν διαφορετικών λογιών απόβλητα, αλήθεια είναι αυτό, αλλά προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα ορίζοντας στόχους ε, και διαφορετικές κατηγορίες αποβλήτων και διαφορετικά μοντέλα για τι επιχειρήσει. Είναι πραγματικά συναρπαστικό να δει κανεί πόσο συμπατικέ βιομηχανίε χρησιμοποιούν ε, τι αλυσίδε διαχείριση των απορριμμάτων και των αποβλήτων ή πώς οι νέε εταιρείε που ξεκινούν την παραγωγή του χρησιμοποιούν την ήδη υπάρχουσα γραμμή τη πρώτη εταιρεία όσο είναι θηγατρικέ, α πούμε. Αυτό θα είναι το μελλοντικό επιχειρηματικό μας μοντέλο, το μοντέλο για τι εταιρείε έτσι κι αλλιώ. Θα έλεγα να σταματήσω εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και τις απόψεις σας, αλλά και τις ερωτήσεις σας. Να συνεχίσουμε το διάλογό μας. Είναι πολύτιμος και για μας να... Είναι σημαντικό να ακούμε τις προτεραιότητες των μελών της Επιτροπής σας. Uh, Ευχαριστούμε θερμά κύριε Αντιπρόεδρε Κατάινεν για την παρουσία σας ε, στην Επιτροπή μας και για την πολύ χρήσιμη παρουσίαση που μας κάνατε και τις ε, Πλήρης και μεστές απαντήσεις που δώσατε. Ευχαριστούμε και προσβλέπουμε σε συνέχιση αυτού του διαρθρωμένου διαλόγου και στο μέλλον.